Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα συνεχίσουμε με το σημείο 9 της σημερινής διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, ΕΤΣΑ, τον κύριο Γκέρτ Ντάντσεπ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. έχουμε αυτές τις τακτικές ανταλλαγές απόψεων για να πληροφορηθούμε για την εργασία των διαφόρων αποκεντρωμένων φορέων που μας ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήλθατε. Όταν πήγαμε στο Ελσίνκι στον οργανισμό σας ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά αυτά που είδαμε και είδαμε και τον ενθουσιασμό με τον οποίο και εσείς και οι συνάδελφοί σας εργάζεστε στα πλαίσια του ΡΙΤΣ για την καταγραφή και την αξιολόγηση όλων των χημικών ουσιών. Τα χρόνια 2007 <clears throat> και μέχρι 2011 ήταν πολύ σημαντικά μέσα στα πλαίσια του προγράμματος αυτού και είναι πολύ σημαντικό που έρχεστε ενώπιον της Επιτροπής μας να μας παρουσιάσετε το έργο σας και θα σας δώσω τον λόγο και μετά θα ακολουθήσει η ανταλλαγή απόψεων. Έχετε τον λόγο. Danke. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, είναι μεγάλη η τιμή για μένα να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσω για, τα, για την υπηρεσία χημικών στο Ελσίνκι για να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας θα ήθελα να τονίσω πέντε σημαντικά θέματα και δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες για τις διάφορες δραστηριότητες ε, της υπηρεσίας μας ε, μέσα στα πλαίσια των κανονισμών REACH και CLP. Και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Καταρχάς ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω για, την, για τις θετικές εξελίξεις σχετικά με το REACH. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία αυτή για μας ε, που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον, ε, και τους πολίτες και το περιβάλλον ε, από τις ενδυνάμει ε, επικίνδυνες και επιβλαβεί συνέπειες των χημικών. Τις επόμενες τρεις εβδομάδες οι περισσότερο επικίνδυνες ουσίες και αυτές οι οποίες παράγονται στις μεγαλύτερες ποσότητες όλη την Ευρώπη θα έχουν καταχωρηθεί στο Ελσίνκι. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Ε, μέσα σε λιγότερο από δυόμιση χρόνια από την ε, στιγμή που μπήκε σε λειτουργία το REACH και ενώ ακόμα προσλαμβάνουμε κόσμο, το προσωπικό του έτσα ε, στο Ελσίνκι έχει καταφέρει να προχωρήσει με αυτή τη διαδικασία με ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματικότητα. Αυτό οφείλεται σε ένα προσεκτικό σχεδιασμό, προετοιμασία, σε συστήματα υποστήριξης και στην πολύ σκληρή δουλειά των συναδέλφων μου. Είμαι πολύ ευτυχής ε, και αισθάνομαι, αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ε, προείσταμε μιας ε, τέτοιας ομάδας αταλαντούχων ε, ατόμων. Από χτες η ΕΤΣΑ έχει δεχτεί μέχρι το 2010 14.015 φακέλους καταχώρησης και έχει εκχωρήσει 10.200 νούμερα καταχώρησης, ε, το οποίο καλύπτει 2.446 ουσίες. Επίσης αυτό δείχνει τον, είναι ένας δείκτης ε, της ε, καινοτόμας δυναμικότητας του, της χημικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε δεχτεί καταχωρήσεις για 834 νέες ουσίες το 94,4% των καταχωρήσεων του 2000 των εγγραφών για το 2010 προέρχονται από μεγάλες επιχειρήσεις, το 4% από μεσαίες επιχειρήσεις και το 1,4% από μικρές. Επίσης έχουμε δεχτεί 550.000 κοινοποιήσεις για την ταξινόμηση και την σήμανση χημικών. Η προθεσμία για τις κοινοποιήσεις για το CLP ε, ε, εκπίπτουν στις 3 ε, Ιανουαρίου του 2011. Γι' αυτό περιμένουμε αρκετά εκατομμύρια υποβολών στην υπηρεσία. Οι διαδικασίες REACH και CLP επομένως έχουν ευτεθεί σε τροχιά και η, η μηχανή της υπηρεσίας μας ε, έχει τεθεί σε λειτουργία. Άλλες περιοχές του κόσμου ε, παρακολουθούν με προσοχή τα τεκτενόμενα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την πολιτική για τα χημικά και μας έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους περιοχές, αρχές του, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, με τις οποίες είμαστε σε στενή επαφή. Ε, υπεύθυνη για αυτή την επιτυχία είναι η προσέγγιση την οποία έχουμε υιοθετήσει. Θέλουμε να δουλεύουμε ανοιχτά και διάφανα. Η... Οφείλω να ομολογήσω ότι όσοι συνεργάζονται μαζί μας έχουν ε, παίξει σημαντικό ρόλο γιατί συμμετέχουν στις συναντήσεις των επιτροπών, μας βοηθάνε ε, και προετοιμάζουν τις επιχειρήσεις η πιο σημαντική καινοτομία που είναι μοναδική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να επιτρέπει στους ε, εμπλεκομένους και σε αυτούς όπου ε, ασχολούνται με τις διάφορες υποθέσεις, να συμμετέχουν με τους διάφορους φακέλους, να συμμετέχουν ε, στις συζητήσεις της Επιτροπής των Κρατών Μελών όταν συζητώνται προτάσεις για δοκιμές στα ζώα. Θα ήθελα να έρθω τώρα σε μια δεύτερη παρατήρηση, σε ένα δεύτερο σημείο. Ποια είναι η προσέγγισή μας για το τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε μια σαφή αποστολή να παίξουμε το ρόλο μας στην εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP, διαχειριζόμενοι τις διαδικασίες σαν κεντρική υπηρεσία και ε, υλοποιώντας συγκεκριμένα καθήκοντα στα, στα ετήσια και στα πολυετή προγράμματα εργασίας, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στο website μας και τα οποία σας έχω στείλει ούτως ή άλλως πριν από τη σημερινή συνεδρίαση, θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες ο, ε, το Ρίτσο, ο, Ρίτσο, ο κανονισμός Ρίτσο είναι ο πιο αυστηρός ε, κανονισμός ε, για τα χημικά σε όλο τον κόσμο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και οι επιχειρήσεις κάνουν τα πάντα για να τον σεβαστούν. ακούμε τις απόψεις της βιομηχανίας και απαντούμε στα θέματα τα οποία τίθενται αναπτύσσοντας πρακτικές λύσεις μέσα, στα πλαίσια, μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο και ε, υλοποιώντα ε, κάποια μέτρα υποστήριξη ε, τα οποία δεν προβλεπόντουσαν ε, στο σχεδιασμό της υπηρεσίας. επίση, Η, επίσης, η εργασία για το DCG είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στις αρχές και στην βιομηχανία για να μπορέσουμε να βρούμε και να ελέγξουμε λύσεις μέσα σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Φέτος για πρώτη φορά κάναμε μια έρευνα και ε, ανάμεσα σε όλους τους ε, εμπλεκομένους και χίλια από αυτοί μας απήντησαν. Στην, σε απάντηση των όσων μας υπέβαλαν έχουμε αυξήσει την υποστήριξή μας και την βοήθεια που προσφέρουμε στην βιομηχανία και όλες αυτές τις ε, συμπληρωματικές πληροφορίες και υπηρεσίες τις προσφέρουμε προς τους συνεργάτες μας γιατί συνεργαζόμενοι μαζί τους και ακούγοντας τους συνεργάτες μας είμαστε αποφασισμένοι να, να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και κάποιες προκλήσεις οι οποίες παραμένουν και θα ήθελα να τις αναφέρω εν συντομία. Τέσσερις από αυτές τις προκλήσεις σχετίζονται με τη διαδικασία καταχώρησης για να απαντήσουμε στις συγκεκριμένες ανάγκες των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων ή για τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ε, κάποιοι χρήστες ε, των χημικών, για το ακαθόδες θέμα της, ε, των δεδομένων που μοιράζονται κάποιες, κάποιες εταιρείες και επίσης για να μειώσουμε δραματικά την, τις επιστημονικές μας δραστηριότητες για να αυξήσουμε συγγνώμη, δραματικά τις ε, βασικές μας επιστημονικές δραστηριότητες σχετικά με τα δεδομένα καταχώρηση και την αξιολόγησή τους μέχρι το 2010 ε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολλές ε, μικρές ε, εταιρείες οι οποίες ασχολούνται και εφαρμόζουν τον REACH. Έχοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά νου, προσπαθούμε να παράγουμε έγγραφα σε 22, στις 22 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε επίσης ε, δημιουργήσει και μία σειρά εγγράφων και fact sheets για να εξηγήσουμε συγκεκριμένα θέματα με έναν πιο συμπυκνωμένο και πιο φιλικό προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τρόπο. Η... Το να μεταφράζουμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το γενικό κοινό κάποια κείμενα και αυτό θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητά μας για να μπορέσουμε να ε, ικανοποιήσουμε τα, τα αιτήματα που υπάρχουν. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για το REACH είναι πώς μπορούμε να μοιραζόμαστε τα δεδομένα και τις ε, πληροφορίες που υπάρχουν. Για να μην, για να μην επαναλαμβάνονται ε, οι δοκιμές ε, στα ζώα που δεν είναι απαραίτητες και για να περιορίσουμε το κόστος για την βιομηχανία, οι κάτοχοι, οι ιδιοκτήτες των δεδομένων για κάποιο χημικό πρέπει να, να τις μοιράζονται με τις άλλες επιχειρήσεις και τους εισαγωγείς. Αυτό δεν ήταν εύκολο ε, με κάποιες επιχειρήσεις ε, οι οποίες αρνήθηκαν να διαθέσουν ε, τα, τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους. Μια άλλη πρόκληση που σχετίζεται με, την, με αυτές τις μεταδεδομένα και το μοίρασμα θέλετε αυτών των δεδομένων είναι ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι δοκιμές, οι χημικές δοκιμές στα ζώα είναι η τελευταία λύση που επιλέγουν οι επιχειρήσεις. Εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά για να είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο στόχος θα γίνει πραγματικότητα. Όλα τα... Οι προτάσεις για τα τεστ που έχουν ε, αξιολογηθεί από την ΕΚΑ έχουν γίνει ομόφωνα δεκτές από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στην Επιτροπή των κρατών μελών ΕΚΑ το οποίο αντικατοπτρίζει θετικά, αν θέλετε, την ανάγκη ε, οι προτάσεις για τις δοκιμές να προωθηθούν στον πιο γρήγορα. Ένα άλλο στοιχείο που αφορά τις εργασίες μας, για να αποφύγουμε ε, μη αναγκαία τεστ στα ζώα είναι η ανάπτυξη διαφόρων εργαλείων που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να καλύψουν τα κενά που έχουν στις ε, πληροφορίες τους συγκρίνοντας τι ουσίε του με κάποιες άλλες ουσίες. Παραδείγματο χάρη η επόμενη ε, εκδοχή του Toolbox XAR του ΩΣΑ ε, θα δημοσιευθεί online. Μια τελική πρόκληση το 2011 είναι να κάνουμε το, με την καλύτερη δυνατή χρήση του πλούτου των πληροφοριών που έχουν προσφέρει οι επιχειρήσεις ε, για, τα, για τις χημικές τους ουσίες ε, με την ε, πρώτη προθεσμία καταχώρησης. Αυτή, αυτές οι πληροφορίες είναι τεχνικής και επιστημονικής φύσης και επομένως αυτούσιες δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές από το γενικό κοινό. Όμως έχουμε δεσμευθεί να τις διαθέσουμε στο κοινό, να είναι προσβάσιμες στο κοινό, έτσι ώστε οι συνεργάτες μας, οι ερευνητές και οι πολίτες που ενδιαφέρονται να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι η τελευταία φάση της, ε, το τελευταίο στάδιο της φάσης δημιουργίας μας ε, εξετάζουμε τις προτεραιότητες που θα πρέπει να υιοθετήσουμε από εδώ και πέρα η επόμενη προθεσμία για, την, ε, για τις αιτήσει καταχώρησης είναι Μάιος του 2013 και στην ενδιάμεση περίοδο θα, θα εστιαστούμε όχι πλέον ε, θα μάλλον θα εστιαστούμε στην επιβολή του REACH στην ε, στον εντοπισμό ενός υψηλότερου αριθμού ουσιών που μας ενδιαφέρουν ε, ε, ιδιαίτερα, substances of very high concern, ε, η επιστημονική αξιολόγηση των καταχωρήσεων και συνεισφορές στην εργασία των νέων επιστημονικών δεδομένων, όπως είναι τα νάνο υλικά και κάποιες άλλες ουσίες που διαταράσσουν την ενδοκρινική λειτουργία. Η εφαρμογή του REACH και του CLP είναι ευθύνη βεβαίως των κρατών μελών και είναι και μια μεγάλη πρόκληση για αυτές. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε βέβαια δίνοντας μια εμπιστευτική πρόσβαση στις πληροφορίες που οι επιχειρήσεις μας προσφέρουν. Ο, ο κατάλογος υποψηφίων για την έγκριση συμπεριλαμβάνει αυτή τη στιγμή 38 ουσίες ιδιαίτερως υψηλού ενδιαφέροντος ε, και άλλες 11 που ε, αυτή τη στιγμή εξετάζονται για να δούμε κατά πόσον θα συμπεριληφθούν. Οι Επίτροποι Ταχάνη και Ποτότσνικ μα είπαν σαφέστατα ποιε είναι οι προσδοκίε μα, οι ότι ο κατάλογο αυτό δηλαδή θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα δύο χρόνια. Τώρα είμαστε στην αρχή τη διαδικασία καταχώρηση και είμαι, σίγουρο ότι ο κατάλογο αυτό θα είναι πολύ διαφορετικό σε λίγα χρόνια. Μία άλλη ε, μεγάλη πρόκληση για το ΕΚΑ τα επόμενα χρόνια είναι να αξιολογήσει τα, τους φακέλους ε, που έχουν ε, υποβάλει οι εταιρείε. Ήδη αναφέρθηκα φακέλους αυτούς ε, αξιολόγησης και στην ε, δουλειά που έχει γίνει για τις προτάσεις σχετικά με τις δοκιμές. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει, ε, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος συμμόρφωσης. Δηλαδή η ΕΚΑ θα πρέπει να εξακριβώνει ότι οι επιχειρήσεις, που έχουν, υποβάλει, ότι οι επιχειρήσεις έχουν υποβάλει φακέλους καλής ποιότητας έχουμε σαν στόχο να πετύχουμε το 5% ελάχιστο 5% αυτών των ελέγχων πριν από την επόμενη προθεσμία καταχωρήσεων ε, το 2013. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ρίτς είναι ένας κανονισμός τελείως καινοτόμος. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε την, ε, ε, την εξέταση, την αξιολόγηση που κάνουμε για τη λειτουργία του Ρίτς και θα υποβάλουμε μέχρι τα μέσα του 2011 την έκθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης η ΕΚΑ θα πρέπει να παρακολουθήσει τα αιτήματα της Επιτροπής για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης στα χημικά και στον ΟΣΕ και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και τώρα στο τελευταίο, η τελευταία παρατηρήση που θα ήθελα να κάνω και αφορά του τομεί που μπορείτε να μα βοηθήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Κοινοβούλιο για τη δουλειά που είχε κάνει τα τελευταία χρόνια, για τον βασικό ρόλο σα ε, στην γέννηση αυτή τη μοναδική ε, νομοθεσία, ε, για την υποστήριξή σα για την εξαιρετική και απρόβλεπτη προσωρινή επιχορήγηση για το ΕΚΑ το 2010. Σε προσωπικό επίπεδο χαιρόμαστε που μπορούμε να μπορέσαμε να καλωσορίσουμε την αντιπροσωπεία της Επιτροπής σας στο Ελσίνκι τον Απρίλιο και, στο Διοικητικό, το Διοικητικό Συμβούλιο εμπλουτίστηκε από τη συμμετοχή του πρώην ε, ε, εισηγητή για το Ρίτσο, του Μπουίντο Σακόνη και του συνεισηγητή του Χάρμουτ Νάσαουερ. Θα ήθελα να σας πω ότι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε μέσα στο πνεύμα του Ρίτσι και του CLP. Το, το πνεύμα αυτό συνεχίζει να ζει, είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, όπως επίσης και η υποστήριξη της καινοτομίας. Θα ήθελα να σας ζητήσω να χρησιμοποιήσετε και την ε, επιρροή σας σε εθνικό επίπεδο. Ο κανονισμός REACH βασίζεται σε μια στενή συνεργασία ανάμεσα στο εθνικό και στο κοινοτικό επίπεδο. Ο ρόλος των κρατών μελών είναι ζωτική σημασία, όχι μόνο για την υποστήριξη της βιομηχανίας μας, αλλά και για την εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και για την ε, και για την ίδια την επιστημονική, τις ίδιες επιστημονικές αποφάσεις. Όλες οι επιτροπές ΕΚΑ ε, συνίστανται από εκπροσώπους και εμπειρογνώμενες των κρατών μελών και η δουλειά της, των εισηγητών της Επιτροπής ε, είναι ουσιαστική για την ποιότητα των ε, αποτελεσμάτων της ΕΚΑ. Κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να σας ζητήσω να μας βοηθήσετε να ευαισθητοποιήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως στην εκλογική σας περιφέρεια. Εάν μπορείτε να το κάνετε να έρθείτε σε επαφή μαζί μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προθεσμία κοινοποίηση ε, του CLP που λήγει στις 3 Ιανουαρίου του 2011 και που εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ποσότητα επικίνδυνης ουσίας που επηρεάζει επομένως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, εμείς στο ΕΚΑ είμαστε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουμε για το ρίτσι και ξέρουμε πώς λειτουργεί πρακτικά. Κανείς άλλος δεν έχει την απαραίτητη γνώση όπως οι συνάδελφοί μου. Και να μας χρησιμοποιήσετε. Παρακολούθησα τις συζητήσεις ε, για την νομοθεσία για ε, τα biocides και εγώ και οι συνάδελφοί μου είμαστε περήφανοι που είδαμε ότι εσείς προτείνατε ε, για τα βιοκτώνα ε, η υπηρεσία μας να έχει έναν πιο ε, έντονο και πιο σημαντικό ρόλο. Και για τα πραγματικά με τη βοήθειά σας ε, τα βιοκτώνα πιστεύω ότι θα ε, έχουν μια πολύ καλύτερη, η νομοθεσία φυσικά, θα έχουν μια πολύ καλύτερη ευκαιρία επιτυχούς εφαρμογής. Περιμένω το τηλέφωνό σας αναλαμβάνω την ευθύνη για το δίκτυο των ε, διευθυντών των υπηρεσιών το Μάρτιο του 2011 ε, και θα ήθελα να σας ζητήσω ε, να χρησιμοποιήσετε τις, την εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις των διαφόρων υπηρεσιών. Πρόεδρε, κύριε Λάινεν, κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να μιλήσω εδώ και περιμένω και τις δικές σας συνεισφορές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντάνσετ για την εισαγωγή αυτή που μας κάνατε και θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων. Όπως σας είπα μας εξέπληξε ήδη το έργο σας στο Ελσίνσχη 750.000 ουσίες οι οποίες πρέπει να ταξινομηθούν Σαράντα ή πέντε ουσίες οι οποίες έχουν καταγραφεί μέχρι τον Νοέμβριο και φυσικά είναι γνωστό το όνομα του Γκίντο Σακόνη Θέλουμε να χαιρετήσουμε και επίσημα και εγκάρδια τον Γκίντο Σακόνη ο οποίος ήταν ο εισηγητής μας για το Ρίτς. Καλώς ήρθες. Και φυσικά μπορείτε να λάβετε και το λόγο εφόσον το επιθυμείτε. Έχουμε και ένα άτομο που είναι ο εισηγητή μα, μάλλον το άτομο επαφή για το Ελσίνκι, που είναι η Σάτου Χάση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θέλω ευχαριστώ τον κύριο Ντάρσετ που ήρθε να συζητήσει μαζί μα. Δύο σύντομα σημεία για τα βιοκτώνα μονάχα και την νομοθεσία που τα αφορά, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην νομοθετική διαδικασία και μερικές σύντομες παρατηρήσεις για το REACH. Όπω ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμπληρώσει την πρώτη ανάγνωση του νομοθετήματος για τα βιοκτώνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρχει μία, ε, σε δύο φάσεις διαδικασία έγκρισης μέχρι το 2015 και το 2017 αντιστοίχως και επίσης αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην υπάρχει το τέλος αυτό το οποίο συνδέεται με την αίτηση έγκρισης το οποίο είναι και μια σημαντική πηγή εσόδων για τον φορέα σας. Μπορείτε να μας πείτε πώς το ατενίζει το θέμα αυτό το, το έτσα, το φορέας για τις χημικές ουσίες, πώς θα επηρεάσει το έργο σας στην πραγματικότητα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε να υπάρχει ένα πιο συντομευμένο χρονοδιάγραμμα για την ε, αξιολόγηση <clears throat> βιοκτώνων προϊόντων αντί για 9 μήνες να είναι 3 μήνες αυτή η προθεσμία. Ποια είναι η απόψή σας τώρα για αυτή την ε, ρύθμιση και το τι θα σημαίνει στην πράξη. Δύο ακόμα σημεία για το REACH. Ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκε στο παρελθόν και που συζητάτε ακόμα τώρα είναι το κατόφλι 0,1% για τις ουσίες οι οποίες βρίσκονται σε, διάφορες, ε, ε, σε διάφορα υλικά και μιλάμε φυσικά για ουσίες οι οποίες θεωρούνται επικίνδυνες και είναι ουσίες που προκαλούν ενδεχομένω κινδύνους. Το 0,1% σημαίνει το σύνολο του προϊόντος. Άμα έχουμε να κάνουμε με μεγάλα αντικείμενα, μεγάλα προϊόντα, όπως είναι τα έπιπλα. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει μια πολύ υψηλή συγκέντρωση τοξικών ουσιών, παραδείγματος χάρη στα εξωτερικά, στις εξωτερικές επιφάνειες ενός επίπλου. Θα ήθελα να έχω την άποψη του φορέα για τις χημικές ουσίες για κάτι τέτοιο, για τα ζητήματα αυτά. Τελευταία μου <clears throat> παρουσίες, η παρατήρηση αφορά τις νανοουσίες. Όπως γνωρίζουμε όλοι υπάρχει μια συζήτηση η οποία εκτελήσεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με το αν το REACH είναι σε θέση να καλύψει τα θέματα ασφάλειας που συνδέονται με τις νανοουσίες ή όχι. Θα ήθελα να ξέρω πόσο φορέα σας λοιπόν αντιμετωπίζει αυτό το θέμα, τι κάνει η ΕΤΣΑ για να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία θα εξασφαλίσει ότι θα δίδονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα νανοηλικά. Και κατά πόσο αυτό το πράγμα είναι ένα θέμα για σας όταν εξετάζετε τους φακέλους οι οποίοι έχουν υποβληθεί προς καταχώρηση και προς εγγραφή. Ευχαριστώ σα του ο Ρίχαρτ Ζέμπερ, όχι Βέμπερ αλλά Ζέμπερ. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάνσερτ για το γεγονός ότι ήρθε ενώπιον της Επιτροπής μας υπάρχει αυτή η σημαντική ημερομηνία του Νοεμβρίου που αναφέρθηκε και είναι απαραίτητο να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν το, η εφαρμογή του REACH που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα νομοθετικά πακέτα που χρειαστήκε να αντιμετωπίσουμε. Ανέφερε ο κύριος ε, Διευθυντής ότι και τον επόμενο χρόνο θα υπάρχουν πολλά θέματα που θα εμπλέκουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταγραφές από μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ένα ερώτημα που θέλω να θέσω είναι ότι πολλές φορές όλη η τεκμηρίωση για τα θέματα αυτά του Ρίτς είναι στα αγγλικά. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε από ένα επιχειρηματία πραγματικά στη Βαυαρία να καταλαβαίνει όλα αυτά τα τεχνικά στοιχεία στα αγγλικά. Μήπως λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει κάποια ρύθμιση που να εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται όλες οι γλώσσες, γιατί ιδίω οι επιχειρηματίε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα έχουν δυσκολία να ανταποκριθούν στι ανάγκε αυτέ τι γλωσσικές. Επίση άκουσα αυτά που είπατε με τι εμπειρίε σα ότι αυτή η πρώτη διαδικασία <clears throat> καταγραφή θα αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο μια σειρμαγιά για τη συνέχεια και θα σας βοηθήσει να καταλάβετε ποια είναι τα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσει. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε ήδη ορισμένε ήδη κάποιες σκέψεις για το τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή την πρώτη διαδικασία καταγραφή ώστε να μπορέσετε να αντιδράσετε με ταχύτερο τρόπο στι μεταγενέστερε καταγραφέ και να οργανωθείτε καλύτερα. Δεν ξέρω λοιπόν πώς θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ε, πληροφορίες. Και εμείς θα θέλαμε από τη δική μας πλευρά να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την ομάδα επαφής των διευθυντών που αναφέρατε εσείς, αν είναι πράγματι ένα χρήσιμο εργαλείο και αν το θεωρείτε εσείς πρόσφορο. Θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας. και κατά πόσο θα δημιουργηθούν και άλλοι φορείς. Έχουμε ακούσει και επίση για το ΣΥΦ ορισμένες διαματήριες, αυτό το φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και πάλι από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα μπορέσετε εσείς να διευκολύνετε το έργο αυτών των επιχειρήσεων που πολλές φορές μπορεί να φαίνεται ότι οδηγεί σε δυσκολίες λόγω της ε, το όγκο των πληροφοριών που πρέπει να δοθεί. Ευχαριστώ, Ρίχαρτ, η Ντάγμαρ, το Ρότ και Μπέρεντ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θυμάμαι ότι πριν από τέσσερα χρόνια βρισκόμασταν σε αυτήν την ίδια αίθουσα και ήταν ο Γκίντο, ο Γκίντο με τους ε, συνεργάτες του και συζητούσαμε για τα θέματα αυτά. Και τότε όλο το σύστημα αυτό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χημικών Ουσιών, η ΕΚΑ, υπήρχε μονάχα στο χαρτί. Και πρέπει να σας πω συγχαρητήρια, με μεγάλο θαυμασμό χαιρετίζουμε τη δημιουργία και τη λειτουργία αυτού του φορέα και πρέπει να σας συγχαρώ και εσάς και τους συνεργάτες σας και αν θέλετε μπορείτε να μεταφέρετε στο Ελσίνκι αυτό το μήνυμα. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Κυρίως αυτό το τελευταίο σημείο που ανέφερε η κυρία Χάση για την ανοτεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην νομοθεσία για τα καλλιντικά και θα παίξει και σημαντικό ρόλο και σε νομοθεσία ασφάλειας τροφίμων κτλ. Το θέμα της ανατεχνολογίας, Επομένω όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή. Πρέπει να μιλήσω και για την ευζοία των ζώων και τις δοκιμασίες σε ζώα. Άκουσα αυτά που είπατε και ήμουν πολύ ικανοποιημένη από αυτά που άκουσα από εσά. Ξέρω ότι προσπαθείτε να κάνετε τα πράγματα διαφορετικά και να έχετε μία αντιμετώπιση που να εξαλείψει το βαθμό του δυνατό της δοκιμασίας στα ζώα χωρίς να μειώνεται το επίπεδο ασφαλείας. Άκουσα επίσης αυτό που είπατε με τον, για τη συνεργασία με τον ΩΣΑ. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθούμε με τον ΩΣΑ, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αλλά ο ΩΣΑ είναι ένας από τους σημαντικούς φορείς μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πώς μπορείτε να πείσετε ένα τέτοιο παλιό οργανισμό να λειτουργεί με σύγχρονους ρυθμούς που είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αν θέλουμε να εξαλείψουμε τις δοκιμασίες σε ζώα. Διαφάνεια. Μίλησατε για τη διαφάνεια και εγώ εκτιμώ αυτά που λέτε. Ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε σε πολλούς φορείς είναι το θέμα της ανεξαρτησίας των εμπειρογνωμών. Η ανεξαρτησία είναι μια μεγάλη λέξη. Είναι δύσκολο να πει κανείς ποιος είναι λευκός, ποιος είναι μαύρος, ποιος είναι γκρίζος. Αλλά τελικά η αλήθεια θα πρέπει να βρίσκεται στα μάτια του έξω κόσμου, αυτών οι οποίοι παρακολουθούν τα θέματα αυτά. Και πραγματικά η αξιοπιστία ενός φορέα εξαρτάται από το πώς την ατενίζουν αυτοί που είναι απ' έξω. Θα ήθελα λοιπόν να έχω μια σαφήνεια για σας, τι ακριβώς σημαίνει για σας η διαφάνεια και η ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι χρησιμοποιούνται για το έργο του φορέα σας και που φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι ο φορέας σας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ε, πολιτών της Ευρώπης. Μπορούμε φυσικά να σας πάρουμε τηλέφωνο αν θέλετε, αλλά ανέφερε και ο κύριος ε, Ζέμπερ σε κάτι το οποίο μπορεί να, ήταν, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο, να έχουμε ένα εύληπτο τρόπο πληροφόρησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα δίναμε στη χώρα μας. Και επίσης, επειδή είμαστε έξι εβδομάδες μοναχά από τα Χριστούγεννα, αν ο Άι Βασίλης σας ζητούσε να του δω, αν μάλλον ο Βασίλης Βασίλης σας ζητούσε να διαλέξει ένα δώρο, τι δώρο θα θέλατε να σας κάνει. Α, ενδιαφέρον αυτό λέω. Ο Chris Davis. Εσύ τι θέλεις για Χριστούγεννα. Εμείς ακούμε να υπάρχουν επικρίσεις από τις ομάδες πίεσης της βιομηχανίας για το ρίσκο και για τον φορέα σας. Είναι καλό να ακούμε λοιπόν αυτή την δήλωση εμπιστοσύνη στο έργο της, ε, του φορέα σας. Πρέπει να συγχαρώ και εσάς και το προσωπικό σας λοιπόν για την ε, προσήλωσή σας στην ε, εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας στην πράξη. Για να επανέλθω όμως στις επικρίσεις. Υπάρχουν οι επικρίσεις αυτές καθυστερήσεις, υπερβολικός όγκος εργασίας που καθυστερεί τα πράγματα, πολυπλοκότητα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για σας, ποια είναι τα κύρια στοιχεία ε, ανησυχίας της βιομηχανίας σε σχέση με το φορέα σας και το ΡΙΣ. Ποια είναι τα θέματα τα οποία θεωρείτε ότι πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπιστούν από σας. Πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Ο Ντάνι Γιώργενσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να επικροτήσω όλα αυτά τα θετικά πράγματα που είπαν οι συνάδελφοι. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το να δούμε ότι κάτι το οποίο ήταν μονάχα άσκηση χάρτου πριν από λίγα χρόνια, τώρα πια είναι ένας πραγματικός οργανισμός με σάρκα και ωστά. Ένα ερώτημα για το REACH μονάχα και κάποια ερωτήματα για τα βιοκτώνα, για το REACH. Και αυτό συνδέεται με αυτό που είπε η Dagmar που είναι οι δοκιμασίες σε ζώα και οι δυνατότητες που υπάρχουν για εναλλακτικέ δοκιμασίες. Και ιδίω σε ό,τι αφορά τη συνεργασία και με τον ΩΣΑ. Γιατί εγώ πήγα στην ΕΚΜΑ, στον δεσμό αυτών και μίλησα με τους εμπειρογνώμονες στην ΙΣΠΡΑ επίσης και είναι ενδιαφέρον πόσο πολλές εναλλακτικέ δυνατότητες υπάρχουν και έχουν θεωρηθεί έγκυρες. Αν δείτε τον αριθμό των ζώων που μπορούν να διαζωθούν με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια ιστορία επιτυχίας, αλλά δεν εφαρμόζεται γενικά. Έχετε λοιπόν μια ευρωπαϊκή διαδικασία εγκυροποίησης των εναλλακτικών λύσεων που θα σώσει τις ζωές χιλιάδων ζώων κάθε χρόνο, αλλά δεν εφαρμόζονται αυτές οι πρακτικές γιατί εμπλέκονται όλα αυτά και στο πλαίσιο του όσα από ό,τι καταλαβαίνω. Μήπως λοιπόν θέλετε να σχολιάσετε αυτό το θέμα και να μας πείτε κατά πόσο τροχοπεδεί την εφαρμογή αυτή η όσα και επίσης γιατί είναι απαραίτητη αυτή η σύνδεση με τον όσα εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει εμεί να έχουμε κάποια σχέση με τον όσα στα θέματα αυτά. Διοκτώνα. Εγώ είμαι γενικό εισηγητή από την ομάδα, το, είμαι μάλλον ο σκιώδη εισηγητή των Σοσιαλιστών για αυτό το θέμα. Και πρέπει να πω ότι έχω νιώσει μια γενικότερη ματέωση για όλη αυτή τη διαδικασία γιατί δεν ήμουν σε θέση να κατανοήσω ποια ακριβώς είναι η άποψη της ECHA ε του φορέα για τις χημικές ουσίες. Ίσως θα έπρεπε να σας είχα ρωτήσει προηγουμένως, αλλά είχαμε αντικρουόμενες πληροφορίες για τα θέματα αυτά. Υπάρχει μια επιστροφή που στείλατε εσείς στην Επιτροπή Αναφερόμενο σε πράγματα που υπάρχουν στο παρελθόν θα ήταν πολύ χρήσιμο μπορείτε να μας πείτε εκπεφρασμένα και ευθαρσώς τι πιστεύετε για τα θέματα αυτά ως φορέας και δεν ξέρω αν εγώ μπορώ να σας προσκαλέσω ή ο εισηγητής ή ο πρόεδρος της Επιτροπής μας αλλά νομίζω ότι όταν περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση και πρέπει να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις θα είναι καλό να είσαστε παρόν γιατί για τις συμβαστικές αυτές λύσεις που θα πρέπει να δημιουργήσουμε. Υπάρχουν σημεία που διαφωνούμε ακόμα και ένα από αυτά είναι πόση πίεση θα πρέπει να ασκηθεί στο φορέα σας. Κανείς δεν έχει καμία ιδεολογική θέση για τα θέματα αυτά, απλώς θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα του φορέα αυτού. Αν μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε και κάποια εκτίμηση για το πόσε ουσίες εμπλέκονται αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό ήταν δύσκολο να μπορέσουμε να το διακριβώσουμε ήδη μόνοι μας. Και επίσης, τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα σε σχέση με τη χρηματοδότηση που θα απαιτηθεί για να μπορέσετε να καλύψετε όλες αυτές τις απαιτήσεις που διατυπώνονται από, από μας και αν υπάρχει πραγματικά ένα κίνδυνος συμφόρησης, έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού κτλ. Και πραγματικά όλα αυτά εξαρτώνται από τον αριθμό των ουσιών που θα πρέπει να αναλύσετε. Εμείς δεν ξέρουμε καν πόσες είναι αυτές οι ουσίες. Βλέπετε αυτή η Επιτροπή νοιάζεται πάρα πολύ. Σας σκέπτεται εσάς, το προσωπικό σας, τα χρήματά σας. Και το να μην σας υπερφορτώσει. Αυτό ήταν και αντικείμενο μιας ευρείας συζήτησης εδώ. Αν μπορώ να κάνω αυτό το σχόλιο, ξέρουμε ότι η Κομισιόν ήταν λιγάκι επιφυλακτική για τα θέματα αυτά, με το να σας δώσει περισσότερο έργο, περισσότερη εργασία, αλλά από την άλλη μεριά είχαμε την συζήτηση για τα βιοκτώνα που μας έχει καθυστερήσει η διαδικασία αυτή εγκρίσεων από 27 κυβερνήσεις και θα πρέπει να επιλέξουμε αν θα υπάρχει μια ευρωπαϊκή διαδικασία έγκρισης. Φυσικά αυτό θα απαιτήσει περισσότερη χρηματοδότηση και περισσότερο προσωπικό. Γι' αυτό θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε μια πολιτική επιλογή αν είναι προς την κατεύθυνση να αναλάβετε τα θέματα αυτά. Μακίνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Διευθυντή για την πάρα πολύ θετική του παρουσίαση και εγώ ήμουνα από αυτούς που πήγε στην ΕΚΑ. Νομίζω ότι ήταν πολύ θετική. Είναι τρομακτικό το έργο το οποίο πρέπει να φέρετε σε πέρας. Έχω κάποιες παρατηρήσεις και μετά ερωτήσεις. Χωρίς τώρα να προδικάσω την αξιολόγηση που θα κάνετε του χρόνου, μπορείτε να μου πείτε τώρα πού βλέπετε να υπάρχουν προβλήματα στην νομοθεσία REACH, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Θέλουμε όλοι να έχουμε καλύτερη ρύθμιση, καλύτερη νομοθεσία. Θα ήταν χρήσιμο αν μας δώσετε κάποιες ενδείξεις τη στιγμή που όλοι μας προσπαθούμε σε πάρα πολλά επίπεδα να ε, διαμορφώσουμε την νομοθεσία. Επίσης για τη χρηματοδότηση του φορέα σας, της ΕΚΑ ένα από τα θέματα που ενδιαφέρει τη βιομηχανία είναι το κόστος το οποίο εμπλέκεται, έχετε ουσιαστικά ένα μονοπόλιο. Δεν υπάρχει άλλος ο οποίος μπορεί να εργαστεί με, τους, με τις βιομηχανίες. Πώς θα μπορούσατε να αξιολογήσετε τη σχέση κόστους ωφέλειας για τις υπηρεσίες σας. Έχουμε συλλέξει πάρα πολλές πληροφορίες και κάνουμε καινοτόμα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά τα θέματα των χημικών ουσιών. Αλλά υπάρχει κάποια ανησυχία από τη δική σας πλευρά ότι ίσω αυτέ οι πληροφορίε μπορεί να μην είναι χρήσιμε. Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στον όγκο τη λεγόμενη πληροφορία και τη αποτελεσματικότητα των ελέγχων που κάνετε και τη αξιολόγηση. Και μα δώσατε ορισμένε ε, προειδοποίησεις προηγουμένω Θα ήθελα να ξέρω και κάποια περισσότερα πράγματα για το θέμα των κρατών μελών και για το πώ θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη. Εάν υπάρχουν γενικά περικοπές στους δημόσιους προϋπολογισμούς και τους πόρους στον τομέα αυτό, που είναι εξάλλου ένας σχετικά καινοφανής τομής, πώς, θα, πώς πιστεύετε πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Ίσως όμως αυτό που είπε και η Ντάγμα προηγουμένω, θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ένα φυλάδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκλογικέ εκλογικές μας περιφέρειες. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ένα εύληπτο τρόπο πληροφόρησης των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και τέλος για την ανοτεχνολογία. Εγώ φοβάμαι ότι προπορεύεται πολύ η τεχνολογία της νομοθεσίας και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις για το πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Και επίσης νομίζω ότι είναι χρήσιμο εφόσον βρεθήκαμε στην ΕΚΑ στο Ελσίνκι να κρατήσουμε την επαφή με μερικούς από τους συναδέλφους σας που ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι και μας βοήθησε. Ίσως λοιπόν πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του πόσα πράγματα μπορούμε να μάθουμε από το φορέα Ευχαριστώ πολύ λέει και ο πρόεδρος ο Χόρστ Σνιαλχάρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πάρει πράγματι πολλές πληροφορίες και στα πλαίσια της εργασίας για το ΡΙΖ είχαμε ήδη τη μέρημνα να μπορέσουμε να δούμε πού θα μπορούσαν να υπάρχουν δυσκολίες με τη βιομηχανία. Νομίζω ότι αυτή τη φορά μπορώ να το το επιβεβαιώσω τι γίνεται, ποιος είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί το τελικό προϊόν και τι ρόλο παίζουν αυτοί οι οποίοι είναι ενδιάμεση κρίκη στην παραγωγή. Και θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε ο Ρίχαρτ Ζέμπερ, ότι το κόστος της μετάφρασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό. Και εμείς έχουμε επαφή με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξέρω πολλές από τη δική μου περιοχή, θα πρέπει να υπάρξει κάποια φροντίδα ώστε να μπορούν να ε, επεξεργάζονται με ταχύτητα τα θέματα αυτά και τους φακέλους χωρίς να υποχρεώνονται να καταφεύγουν πάντα σε μεταφραστές. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι μια τροχοπέδη και ένα προσθέτο κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα τελευταία που είπατε με ενόχλησαν λιγάκι είπατε ότι ο φορέας έχει πολύ μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη. Αυτό το πιστεύω. Και όπως σας κατάλαβα, είπατε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η ικανότητα που έχετε συσσωρεύσει. Αυτό σημαίνει ότι και θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο και η εθνοδηγία των βιοκτώνων. Θα μπορούσε το δικό σας προσωπικό δηλαδή να αναλάβει μια τέτοια αρμοδιότητα. Εάν ναι, τότε θα πρέπει να, εάν όχι, θα πρέπει να πούμε και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ότι πρέπει να ενισχυθούν οι ικανότητες που έχετε στην ε, υπηρεσία σας. Κυρία Μακίουεν, Μακέβαν. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάνσαρτ και το φορέα αυτό, την ΕΚΑ που είναι παρόντες ενώπιόν μας. Είναι πολύ καλό επίσης που είναι παρόν και ο Γκουίντο Σακόνη και είναι χρήσιμο να κρατήσει ένα συνεχή διάλογο με το Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Δύο παρατηρήσεις γενικά για τους αποκεντρωμένους φορείς. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερη σχέση το Κοινοβούλιο με τους αποκεντρωμένους φορείς. Τώρα συναντιόμαστε κάθε τόσο καλό είναι, αλλά αυτό δεν δίνει πάντα απάντηση στα ερωτήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση από τους εκλογείς μας. Και υπάρχει και ένα ευρύτερο θέμα όταν θέλουμε να πάρουμε αποφάσεις ε, νομοθετικού χαρακτήρα. Από τη μια μεριά έχουμε την ε, Επιτροπή που μας λέει αυτό δεν γίνεται, από την άλλη μεριά λέμε, λένε τα λόμπι οπωσδήποτε γίνεται. Είναι καλό να έχουμε και μια τρίτη γνώμη. σίγουρα έχετε μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να διαμορφωθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαζόμαστε να έχουμε ένα ειλικρινή διάλογο μαζί σας θα πρέπει να ξέρουμε όταν νομοθετούμε κάτι αν αυτά τα οποία αποφασίζουμε είναι εφικτά ή αν μπορούν να γίνουν με διαφορετικό τρόπο, μπορούν να βελτιωθούν και πολλές φορές όπως και με τα βιοκτώνα χρησιμοποιούμε μία, ε, ένα νομοθέτημα και μεταφέρουμε τις διατάξεις του σε ένα άλλο νομοθέτημα που αυτό πάντα δεν είναι ε, πρόσφορο. Χαίρομαι λοιπόν για αυτά που είπατε με τις αποκεντρωμένους φορείς. Ξέρω ότι κάποια από αυτά τα θέματα είναι ευαίσθητα και για την Επιτροπή, αλλά εμείς είμαστε οι πρώτοι που παίρνουμε τις διαμαρτυρίες, είσαστε οι πρώτοι οι οποίοι έχετε κάποια συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής. Ένα ερώτημα το οποίο μου έχουν αναφέρει πολλές εταιρείε και ίσως ε, έχω χάσει κάτι που είπατε. Ε, μιλάτε για τους... Ε, κατάντι χρήστες, τους downstream users. Ε, να υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα που να μπορούν να δουν αυτοί τις χρήσεις των προϊόντων που έχουν καταγραφεί. Αλλά ενδεχομένως θα υπάρχει και ένα χρονικό χάσμα, δύο ή τρεις μήνες μεταξύ της 30ης Νοεμβρίου και τη στιγμή που θα έχει κάθε χημική ουσία ένα αριθμό καταγραφής, ένα αριθμό μητρώου. Εγώ κατάλαβα ότι αν δεν έχουν ένα αριθμό μητρώου αυτές οι ουσίες, είναι παράνομο να την χάνουν εμπορία. Οπότε με απασχολεί το πόσο θα διαρκέσει αυτό το χρονικό χάσμα και μπορείτε να δώσετε ε, διαβεβαιώσει τους κατά χρήστες ότι αν δεν, ακόμη και να μην έχουν αυτό τον αριθμό θα μπορούν να συνεχίσουν το εμπόριο αυτών των ουσιών. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Γκουίντο Σακόνη. Αν θέλει να λάβει το λόγο, έχει το λόγο Γκουίντο για την ΕΚΑ. Θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ να διαπιστώσω, διαπιστώνοντας μάλλον, ακούοντας όλους τους προαλαλήσαντες ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Δηλαδή συμμεριζόμαστε μια απόψη, δηλαδή για τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας. Πριν μόλις τέσσερα χρόνια, ήμασταν πολλοί οι οποίοι αρνηθήκαμε να δώσουμε έστω και ένα ευρώ σε αυτό το βουνό θα λέγαμε παραγράφων ε, κειμένων ε, ένα περιεχόμενο το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προσδιορίσει. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τότε ότι θα καταλήγαμε σε αυτό που μας περιέγραψε ο κύριος Τζαν Σέτ σαν μια καινοτόμα προσπάθεια. Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε πλέον πολύ θετικά. Ξέχασα όμως τις ευχαριστίες. Να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή για το Περιβάλλον που με έχουν ε, που έχουν δείξει εμπιστοσύνη τέλος πάντων απέναντί μου. Ε, ε, θα ήθελα να πω ότι ειλικρινά πολεμήσαμε με το Συμβούλιο για να πετύχουμε κάτι και ε, είναι για πρώτη φορά που έχουμε και σαν κοινοβούλιο προσώπηση σε, ένα, σε μια υπηρεσία. Κάτι που δεν γίνεται μόλις στις άλλες. Μια εκπροσώπηση στο Συμβούλιο της υπηρεσίας. Επίσης, να ευχαριστήσω τον κύριο Νταν Σετ για το έργο του. Ένα έργο το οποίο συνεχίζει τώρα, μαζί με τους συνεργάτες του εννοείται, ε, 400 άτομα, δεν κάνω λάθος, με διάφορες αρμοδιότητες υψηλού επίπεδου ε, ικανότητες. Πραγματικά είναι μια καινοτόμως προσπάθεια, κάτι που δεν υπήρξε πριν. Και όλοι αυτοί ήταν σε θέση να μπορέσουν να θέσουν σε εφαρμογή, ε, θα έλεγα, αυτό εδώ το έργο ένα έργο στο οποίο έχουμε μια συσυμφόρεση ε, γνώσεων. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε εδώ με μια ζώνη η οποία ήταν σκοτεινή και τώρα ρίχνουμε το φως. Σε σχέση δηλαδή με όλες αυτές τις ουσίες οι οποίες είναι επικίνδυνες και οι οποίες δεν είχαν εντοπιστεί ε, με καταχώρηση, αξιολόγηση και όλα αυτά. Είναι ε, καμιά φορά ίσως δεν είναι δυνατό αλλά είναι επιθυμητό. Φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες που υπάρχουν, υπήρξαν προβλήματα, μέρα-μέρα ε, χρειαζόταν να κάνει κανείς προσπάθεια για να ξεπεράσει διάφορα προβλήματα. Υπάρχουν επίσης διαδικασίες ε, που μπορούν να εφαρμοστούν και υπάρχουν πάντοτε απρόβλεπτες καταστάσεις. όταν θα φτάσουμε την ημερομηνία της 30 Νοεμβρίου που θα γίνει μαζική καταχώρηση θα ε, έχουμε μια κατάσταση στην οποία σίγουρα δεν θα υπάρχουν πλέον προβλήματα. Τώρα, συνομοθετική διαδικασία. Εδώ είχαμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια της Επιτροπής. Είχαμε να κάνουμε με τη μετατροπή μιας δυνατότητας σε κάτι που θα λέγαμε μια υποχρέωση. Δηλαδή, τα δεδομένα τα οποία να μπορούν να μοιράζονται, να τα έχουν αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να έχουν γνώση. Και αυτό είναι προ συμφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνεργασία με την Βρετανική Προεδρία θέλησε να παρέμβει κυρίω για να μπορέσει να υποστηρίξει και τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι μια επί τη αλλαγή. για να καταλήξει κανείς σε μια θα λέγαμε νομική αρχιτεκτονική ε, και πώς καταλήξαμε σε αυτό και γιατί μιλάω για, για όλα αυτά. Γιατί θα ήθελα εδώ να επιστήσω την προσοχή σας, δηλαδή ότι υπάρχει κάτι ουσιώδες. Το REACH, έχουμε ένα κανονισμό, ο οποίος αποτελεί μια μοναδική εμπειρία ποτέ πριν δεν είχε ξεκινήσει μια τέτοια θα λέγαμε επιχείρηση με αυτό το καταπληκτικό τρόπο. Ακόμα και αν έχουμε δυσκολίες. Αποτελεί μια πρόκληση. Εσείς σαν νομοθέτες θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τις όποιες διορθώσεις. Τότε, ξέρετε, κάποιοι που του έλεγα τελειομανείς δεν ήταν ευχαριστημένοι. Αλλά ίσως να μην ήταν και τόσο άδικη αυτή η προσέγγιση αν είχε προσπαθήσει κανείς να επιδιώξει μόνο το τέλειο, δεν θα μπορούσαμε καν να ξεκινήσουμε. Ακόμα θα συζητούσαμε, η υπηρεσία δεν θα υπήρχε. Ακόμα θα μιλούσαμε. Και θα κλείσω κύριε Πρόεδρε. Ε, συγγνώμη που μακρηγορώ. Ε, δεν έχω τη συνήθεια να μιλάω. Ευρωπαϊκά. Λοιπόν, έχουμε ε, την πρόβλεψη Φερπίν ενός προγράμματος το οποίο θα έχει να κάνει με την επαλήθευση που προβλέπει δυνατότητες μιας αναθεώρησης, συμπληρωματικών ε, διατάξεων κτλ. Και όλα αυτά ε, στα πλαίσια του 2000, με την προοπτική του 2012 δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε εκεί στροφή 160 μοιρών. Θα υπάρχει δυνατότητα να γίνονται προτάσεις νομοθετική φύσεως και να δει κανεί τα πλαίσια της, του πεδίου εφαρμογή ε, του κανονισμού. Και χαίρομαι με όλες τις νίκες που έχουν γίνει ε, από όλες τι πτυχέ. Ε, ξέρετε ότι έχουν να κάνουν και με ουσίε, φέρει που ε, παλιότερα θέλαμε να αποκλείσουμε από το πεδίο εφαρμογή του REACH. Αλλά με αυτά ας κλείσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ Γκουίντο Σακόντι. Πραγματικά δεν είναι δύσκολο να βρει κανεί την ε, άκρη και το μύτο της αριά μέσα από αυτό τον κικαιώνα άρθρων, παραρτημάτων κτλ. Επίσης υπήρξε και ένα θέμα για τα βιοκτώνα στην αντίστοιχη ε, οδηγία ο Καρλ Χάντς Φλόρενς νομίζω ήθελε κάτι να πει παραλίγο να μην τον δω κιόλας αλλά ήθελε να λάβει το λόγο μετά από τα θετικά λόγια που είπε ο Γκουίντο Σακόνη Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που πρέπει και εγώ να τον συγχαρώ για το πολύ καλό έργο το οποίο έφερε σε πέρας. Υπήρχαν ήδη από τότε κριτικές για διάφορα πράγματα, αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα για τις ουσίες που είναι πολύ υψηλής, ε, μας οδηγούν σε πολύ υψηλές φροντίδες όπως λέγεται, 83, τώρα έχουν προσθεθεί ακόμα άλλες 11 τέτοιες ουσίες. Πώς γίνεται τώρα αυτό, με τα κράτη-μέλη και όλα αυτά με τον αριθμό των ε, εργαζομένων που έχετε που είναι συγκεκριμένος και με ένα όγκο εργασίας ο οποίος δεν είναι προβλέψιμος. Πώς θα γίνουν τα πράγματα αν, γίνει, αν διπλασιαστεί ο όγκος εργασίας που έχετε για τις εγκρίσεις. Εγώ άκουσα λοιπόν αυτά που είπε ο Γουίντο Σακώνη, ο οποίος είπε ότι φέρεται σαν να είναι <laughs> το αφεντικό της Ευρώπης. Εσείς έχετε κάποια... Τι σχέση ακριβώς έχετε με την Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Ποια είναι η δική σας εντύπωση. Ε, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε εσείς όλο το έργο αυτό. Χρειάζεστε την προστασία του Κοινοβουλίου και τη βοήθεια. Και επίσης για την έννοια μια ουσία, μια καταχώρηση. Αυτή ήταν μια ρύθμιση η οποία άλλαξε πάρα πολλές φορές και όλα αυτά δεν μας έχουν ε, εμάς ενθουσιάσει ιδιαίτερα. Τι έγινε για τα θέματα αυτά. Γιατί οι βιομηχανικοί κύκλοι είχαν να κάνουν πάρα πολλές, κάναν πολλές κριτικές για τα θέματα αυτά. Φαντάζομαι ότι εσείς θα έχετε μια πιο αντικειμενική εικόνα για όλα αυτά τα θέματα. Εντάξει. Μια, ένα μεγάλο φάσμα από ερωτήσεις και σχόλια. Έχετε το λόγο κύριε Ντάνσερτ για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσπαθώ να ακολουθήσω μια διαδικασία βήμα προς βήμα και να ξεκινήσω πρώτα για τα θέματα που αφορούν το REACH. Καταρχήν, το 0,1 ως κατόφλιο για την παρουσία ορισμένων ουσιών σε ένα προϊόν. Τι είναι ένα προϊόν, αυτό είναι το ερώτημα που θέσατε. Ο ορισμός που χρησιμοποιείται στο REACH και σε άλλα νομοθετήματα είναι διαφορετικός και τουλάχιστον σύμφωνα με την ερμηνεία της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν δεν επιτρέπει μια ερμηνεία ότι ένα προϊόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει ότι απαρτίζεται από ομογενή κομμάτια. Δηλαδή η αρχική διατύπωση ήταν σε ένα προϊόν ή στα ομογενή ε, τμήματα ενός προϊόντου. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό λοιπόν να κοιτάμε τα ομοιογενή συστατικά ενός ε, προϊόντος στην περίπτωση του ρίτσου. αρχική αυτή κοιταμε τα ομογενή συστατικα ενος προιοντος στην περιπτωση είχε 6 με 7 κράτη-μέλη που διαφωνούσαν και είχαν μια διαφορετική ερμηνεία από ό,τι τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη αυτά έχουν ε, έλθει με νέες προτάσεις αναφέροντας ότι δεν πρέπει να δούμε μόναχα το σύνολο, το συνολικό προϊόν αλλά και οποιοδήποτε άλλο προϊόν το οποίο είναι ενσωματωμένο στο περιού ολόγου άρθρο. Μπορεί να του περί ε, προϊόν. Μπορεί να υπάρχει ένα προϊόν το οποίο περιέχει άλλα προϊόντα. Και τότε αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να θεωρούνται ότι παραμένουν προϊόντα ακόμα και όταν έχουν ενσωματωθεί σε ένα ευρύτερο προϊόντο. Όλα αυτά λοιπόν τα κράτη-μέλη νομίζω ότι τα αντιμετωπίσουν θετικά. Ένα μεγάλο αριθμό κρατών υποστηρίζει μια τέτοιου είδου ερμηνεία. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο τα κράτη-μέλη αυτά ζήτησαν από την Κομισιόν να ζητήσει μια νέα γνωμοδότηση σε νομικό επίπεδο και εμείς αυτό ζητήσαμε την Κομισιόν, αλλά από ό,τι το κατανοώ ότι σήμερα, μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει επίσημη αίτηση από την Κομισιόν για νομική γνωμοδότηση. Εμείς όμως μέχρι την 1η Δεκεμβρίου θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Αν θέλουμε να εκδώσουμε νέες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να το πράξουμε μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Εμείς προσπαθούμε πάντα να δίνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές 6 μήνες πριν από την τροποποίηση των ε, κανονισμών του ΡΙΤΣ. Το άρθρο 7 του κανονισμού τίθεται σε εφαρμογή του χρόνου τον Ιούνιο. Θα έπρεπε το ταχύτερο δυνατό το Δεκέμβριο να έχουμε δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για το άρθρο αυτό, το 7. Γι' αυτό εμείς ζητήσαμε τα κρατη να μας ε, δώσουν την έγκρισή τους για τη νέα επαναδιατύπωση των κανονισμών που βασίζεται στην παλιά ερμηνεία, αλλά να ζητήσουμε και την ερμηνεία τους και την νομική γνωμοδότησή τους για την νέα διατύπωση. Αν δεν έχουμε καμία νομική γνωμοδότηση μέσα στις 15 Νοεμβρίου θα πρέπει να βασιστούμε στην παλιά ερμηνεία και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε μια γραπτή διαβούλευση στο Διοικητικό Συμβουλίο μας βάσει των κειμένων πρακτικών μας για τις κατευθυντήρες γραμμές τις οποίες δεν Ένα δεύτερο θέμα είναι το θέμα των νανοηλικών που αναφέρθηκε πολλές φορές. Τα νανοηλικά δεν καλύπτονται χωριστά μέσα στο REACH. Αυτό το οποίο καλύπτεται μέσα στο REACH είναι όλα τα είδη όλες οι μορφές μάλλον οι φυσικές μορφές που μπορεί να πάρει μια συγκεκριμένη χημική ουσία καλύπτονται. Και θα πρέπει να εξετάσουμε πάντα αν κατά όγκο περνούν ένα ορισμένο κατόφλι. Άμα πάρουμε παραγωγικά χάρη τον άνθρακα σε άμορφη μορφή, carbon black, αν πολιθεί σήμερα είτε σε μορφή νανοηλικού είτε σε άλλη μορφή, όλα αυτά καταμετρώνται από κοινού για να ξέρουμε αν είναι πάνω από χιλιτόνι παραγωγή χάρη που είναι το κατόφλι μας ενδιαφέρει στην περίπτωση του άνθρακα. Οπότε οι εταιρείε οι οποίες κάνουν μια έκθεση περί ασφάλειας σε χημικό επίπεδο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατές χρήσεις αυτού του υλικού. Και κάποιες από αυτές τις χρήσεις αφορούν νανοηλικά και όχι απλώς άνθρακα σε φυσιολογική μορφή. Οι χρήσει αυτές λοιπόν θα πρέπει να την χάνουν εκθέσεως σε αυτή την περίπτωση στο φάκελο περί νομοθεσίας. Ένα παράδειγμα θέλω να σας δώσω. Μας ζήτησε και η Κομισιόν να συμπιλήσουμε μια έκθεση μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2011 που να περιλαμβάνει πληροφορίες για τα είδη και τις χρήσεις νανοηλικών που έχουν καταγραφεί μέχρι την πρώτη καταληκτική προθεσμία ώστε να μπορεί η Κομισιόν <clears throat> να κάνει μια έκθεση σας, ακόμα και ένα νοέκθεση. έκθεση. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο της, ε, του προβλήματος. Το άλλο στοιχείο του προβλήματος είναι ότι φυσικά θα πρέπει να αξιολογήσουμε αν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες στον φάκελο που συνοδεύει κάθε υλικό σε σχέση με τις χρήσεις τις οποίες μπορεί να τεθεί. Και εδώ έχουμε μπλέξει με ένα προβλημάτων που έχουμε σε ό,τι αφορά την, τους νανοχρήστες και τις νανοχρήσεις και περιμένουμε ακόμα την νανοαπάντηση της Κομισιόν για τα νομικά αυτά νανοθέματα. Προτού συμπληρώσουμε λοιπόν τον έλεγχο αυτών των φακέλων. Κάτι το οποίο θα πράξουμε μέσα στο γενικό χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους συμμόρφωσης που σας ανέφερα προηγουμένως. σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το πώς τις επηρεάζει το ρίσο και την καταληκτική προθεσμία για την καταγραφή των ουσιών. Εγώ προσπάθησα να σας δώσω ορισμένα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι το ποσοστό καταχώρησης, το ποσοστό εγγραφής που έχει υποβληθεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 5% μονάχα που είναι πολύ λιγότερο από αυτό που είχαμε προηγουμένως ε, προβλέψει. Αυτό σημαίνει ότι ζορίζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να υποβάλουν τους φακέλους καταχώρησης. Και δεν ακριβώς η ομάδα επιχειρήσεων που παίρνει την ε, ηγεσία ενδιαφέρονται περισσότερο για τη διαδικασία κοινή καταγραφής που θα ακολουθήσει και θα υποβάλουν τους φακέλους καταγραφής αναφερόμενοι στην διαδικασία κοινή καταγραφής. Όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τις κατευθυντήριες γραμμές είναι μεταφρασμένα σε όλες τις γλώσσες και αυτό έγινε γέρος. Και έχουμε πολλά ακόμα έγγραφα τα οποία έχουν ε, μεταφραστεί και επίσης και το Reach IT καθώς και ο Ευκλήδης που είναι ηλεκτρονικά εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία είναι καταρχήν στα αγγλικά αλλά υπάρχει και ένα εργαλείο βοήθειας σε άλλες γλώσσες. Κάποιος ο οποίος λοιπόν δεν σκαμπάζει από, τα αγγλικά, μπορεί να κάνει κλικ σε ένα κουτί και θα του αναφέρει στη δική του γλώσσα τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Ούτως πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα δυνατό να κάνει κανείς μια υποβολή και εξάλλου η μόνη εταιρεία η οποία διαμαρτυρήθηκε για το θέμα των γλωσσών και είναι μια γερμανική εταιρεία όπως ε, αναφέρατε και έχει στείλει πολλά γράμματα σε εμά και στην Κομισιόν για τα θέματα τα γλωσσικά, στα γερμανικά φυσικά. Εμείς ήρθαμε σε επαφή με αυτή την ε, εταιρεία και είπαμε έχουμε πέντε Γερμανούς, μπορούμε να σας βοηθήσουμε καθόλου. Και η εταιρεία αυτή έχει ήδη υποβάλλει 10 προτάσεις καταχώρησης και δεν έχει κανένα πρόβλημα με την καταχώρηση αυτή που έγινε, απλώς διαμαρτύρεται για ένα θέμα αρχής. Όλα αυτά δημιουργούν ίσως μια υπερβολική εντύπωση γιατί στην πράξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν καταχωρήσεις. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εκπαιδεύσει όλα τα εθνικά γραφεία βοήθειας που ήταν το εργαλείο το οποίο επέλεξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε ε, εκπαιδεύσει τους αρμοδίους των γραφείων βοήθειας να βοηθούν τις εταιρείε να συμπληρώνουν τα έγγραφα αυτά και να τους βοηθούν με τα γλωσσικά θέματα. Και έχουμε φυσικά και κάποια βίντεο τα οποία είναι υποτιτλισμένα στις εθνικές γλώσσες και εξηγούν πώς γίνεται η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων του ρίσου. και έχουμε ακόμα και δεχτεί την αίτηση της ε, Κομισιόν να εξετάσουμε την αναγκαιότητα περαιτέρω μετάφρασης των ε, εργαλείων μας και της πληροφορικής. Έχουμε ε, επίσης ένα εργαλείο πληροφορικό το οποίο έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες, κάτι το οποίο απαιτούσε πάρα πολύ προσπάθεια. Επομένως, έχουμε στην κάθε γλώσσα στην ιστοσελίδα μας, να εξηγούμε τι είναι αυτά τα οποία έχουν μεταφραστεί και τι όχι. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία είναι ε, εγχειρίδια, εργαλεία βοήθειας, όλα αυτά έχουν μεταφραστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. <clears throat> Είναι σημαντικές βέβαια οι γλώσσες, αλλά δεν αποτελούν ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Κάθε φορά που εμείς προχωρούμε σε επίπεδο δημόσιο με τις πληροφορίες που έχουμε για το CNL, με την ετικετοποίηση και στην ομάδα των διευθυντών έχουμε κάνει τη δημοσίευση μόνο όταν υπάρχουν όλες οι ε, γλώσσες, όλες οι γλωσσικές μορφές διαθέσιμες για να μην δώσουμε ένα πλεονέκτημα σε ορισμένες μοναχά γλωσσικές κοινότητες. Νομίζω λοιπόν ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτή την αίτηση που υπήρξε και από την πλευρά του Επιτρόπου Ταγιάννη και την πήραμε πολύ σοβαρά. Και το επόμενο στοιχείο αφορά την ομάδα επαφής των διευθυντών και το κατά πόσο αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, κατά πόσον αξίζει τον κόπο να διατηρήσουμε αυτή την ομάδα επαφών διευθυντών. Αυτό το οποίο όμως έχουμε εδώ είναι μια ομάδα επαφών η οποία ήταν αυτοτελή σε σχέση με τους σκοπούς που εξυπηρετούσε καταρχήν γιατί η κατάρτιση προηγουμένως δεν λειτουργούσε με τον κατάλληλο τρόπο και η βιομηχανία είχε εντοπίσει ορισμένα θέματα τα οποία δεν καλυπτόντουσαν από την νομοθεσία, δηλαδή εξαιρετικές καταστάσεις, έκτακτες καταστάσεις που θα ήθελαν να βρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπιστούν. Και όταν είχαν συλλεγεί όλα αυτά τα στοιχεία, ήμασταν ήδη στην αρχή του χρόνου και δεν είχαμε ακόμα τη δυνατότητα, δεν είχαμε πια τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με την κανονική διαδικασία κατευθυντήρων γραμμών. Γι' αυτό δημιουργήσαμε και αυτή την ομάδα επαφή των διευθυντών. Η Κομισιόν δέχτηκε να παίξει ένα ηγετικό ρόλο μέσα στην ομάδα αυτή και καταλήξαμε σε ορισμένε προτάσει, καταλήξαμε σε ορισμένε λύσει για όλε αυτέ τι περιπτώσει που έχριζαν ρύθμισης και για τις έκτακτες αυτές καταστάσεις που ήταν φανερό ότι η νομοθεσία δεν κάλυπτε επαρκώς τα προβλήματα αυτά. Το εξηγήσαμε αυτό και στα κράτη-μέλη, τα οποία δεν ήταν τμήμα της διαδικασίας απόφασης και επομένως δεν είχαν υποστήριξη και τις λύσεις, αλλά οι λύσεις υπάρχουν, εφαρμόζονται και η ελπίδα μας είναι ότι οι ελεκτικές αρχές θα δεχτούν αυτές τις λύσεις. Το αν θα συνεχιστεί η ύπαρξη αυτη τη ομάδα επαφή το συζητούμε ακόμα. Αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να αντλήσουμε διδάγματα και έχουμε συμφωνήσει με αυτή την ομάδα να αξιολογήσουμε αυτά τα οποία έχουν γίνει σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη λύσεων και επίσης σε σχέση με τα άλλα ζητήματα τα οποία εμπλέκονται. Δοκιμασίες σε ζώα και όσα. Νομίζω ότι το ΡΙΣ προβλέπει την αποδοχή εναλλακτικών ε, δοκιμασιών ακόμα και όταν δεν υπάρχει μια συμφωνία του ΩΣΑ για όλα αυτά τα θέματα. Υπήρξε μια αλλαγή την τελευταία στιγμή η οποία εισήχθη να μας επιτρέπει όταν υπάρχει ευρωπαϊκή έγκριση για μια νέα δοκιμασία να μπορεί να την χρησιμοποιεί μια εταιρεία. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, εμείς υποστηρίζουμε την Κομισιόν στο έργο το οποίο γίνεται στα πλαίσια του ΟΣΑ για τις μεθόδους δοκιμασίας και δεν είναι εύκολο αυτό το έργο γιατί σε τελική ανάλυση δεν είναι χρήσιμο το να εγκαταλείπουμε μία δοκιμασία αν δεν είμαστε σίγουροι σε επιστημονικό επίπεδο ότι η εναλλακτική διαδικασία δίδει ε, σωστά ότι Εάν κάνουμε ένα λάθος μπορούμε να δημιουργήσουμε καρκίνο στους ανθρώπους Πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι και οι επιστήμονές μας λαμβάνουν πάρα πολύ στα σοβαρά αυτά τα προβλήματα και συμβάλλουν καλή την πίστη και καλή την επιστήμη και με την κατάλληλη υποστήριξη. Βιοκτώνα. Βιοκτώνα. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί ήταν πολλά τα ερωτήματα για τα βιοκτώνα. Πρέπει και εκεί φυσικά να βασιστούμε στην σωστή επιστημονική πρακτική. Το να διατυπώσουμε μια επιστημονική γνώμη σε τρει μήνε, αυτό δυστυχώ δεν μπορούμε να το κάνουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Η Κομισιόν είχε προτείνει εννέα μήνε, το Συμβούλιο ήθελε έξι μήνε. Εμεί θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να, να πόσο, πόσο πιο σύντομος μπορεί να είναι ο χρόνος αν κάνουμε όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική τη διαδικασία στο φως των διδαγμάτων του REACH. Αν μας είχαν ζητήσει τη γνώμη μας όταν έγιναν οι, οι προτάσεις, εμείς θα είχαμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση των προτάσεων. Έχουμε δει Είδαμε το δημοσιονομικό δελτίο μεν από την πλευρά της Κομισιόν, αλλά μετά ακολούθησε πάρα πολλούς χρόνους μέχρι την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η απάντηση της Κομισιόν δεν έγινε μετά από διαβούλευση με εμά μετά την πρώτη σας ανάγνωση. Έκτοτε συνήφθηκε πάλι επαφή με την Κομισιόν, αλλά από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει ακόμα κάποια υπηρεσία στην Κομισιόν η οποία είναι υπεύθυνη για τα βιοκτώνα και εμείς υποστηρίζουμε αυτή τη μονάδα όσο μπορούμε περισσότερο. Αλλά μία από τις κύριες ελλείψεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το γεγονός ότι η πρόταση της Κομισιόν θεωρεί ότι η ΕΚΑ μπορεί μέσα σε 12 μήνες να είναι έτοιμη μετά από τη διατύπωση μιας πρότασης για τα βιοκτώνα. Για το ρίσκο χρειαστήκαμε να προετοιμαστούμε τρία χρόνια για να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Αν θέλετε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και για τα βιοκτώνα όπως κάναμε στο ΡΙΣ, δεν μπορούμε να το κάνουμε σε ένα χρόνο, πρέπει να ξεκινήσουμε και νωρίτερα να προετοιμαζόμαστε. Αυτό είπαμε στην Κομισιόν και γι' αυτό παίρνουν κάποια έκτακτα μέτρα να μας δώσουν και περαιτέρω πόροι χωρίς χρήμα και προσωπικό. Είναι ένα είδος ακροβατικής ώστε θα μας εξασφαλίσει τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε για τα βιοκτώνα. Πάση περιπτώσει έχουμε εμπειρογνώμονε για τα βιοκτώνα και θα αρχίσουμε ήδη να εργαζόμαστε για τα θέματα αυτά και μπορούμε να σα υποστηρίξουμε όταν χρειάζεται τη βοήθειά μα, όπω εξήγησα σήμερα το πρωί και στον εισηγητή σα, ο οποίο δεν μπορούσε να έρθει το απόημα ποια ήταν τα κυριότερα στην εισηγητρία σα ποια ήταν τα κυριότερα σημεία και τα έχει καταγράψει και ξέρει ότι, είναι, ότι είμαστε έτοιμοι να σα βοηθήσουμε σε επίπεδο δεύτερη ανάγνωση. Για τον κατάλογο επιθυμητών ονείων ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει καλά η διαδικασία καταχώρησης και ότι θα μπορέσουμε αυτή τη φάση να την καλύψουμε με γαλήνιο τρόπο και προς το συμφέρον όλες τις βιομηχανίες. Για τα τέλη, ναι, χρειαζόμαστε επαρκή τέλη. Αλλά αν τα τέλη αυτά μπορεί να πάρουν το χαρακτήρα όχι κατά αποκοπήν και τελών υποβολής αλλά ετησίων τελών θα είναι καλύτερο γιατί λόγω της ανάγκης να υπάρχουν κάποια τέλη που καταβάλλονται με την εγγραφή πολλές εταιρείε έχουν αποσυρθεί από την αγορά χωρίς να πληροφορήσουν τους πελάτες τους. Ενώ το Ρίτσι δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Έχουμε πολλά προβλήματα λοιπόν με τους πελάτες οι οποίοι δεν παίρνουν πια απάντηση από τους προμηθευτές τους και τους λένε τώρα ότι ορισμένε χημικές ουσίες δεν θα μπαίνουν στην αγορά γιατί αποφάσισαν ότι το ριτς κοστίζει πάρα πολύ. Εάν λοιπόν το κόστος μπορεί να κατανεμηθεί σε, χρονικό, σε ευρύτερο χρονικό ορίζοντα θα έχουμε ένα πιο εύκολο δρόμο προς το μέλλον και αυτό είναι και το μήνυμά μου για τα βιοκτώνα. Αν πείτε ότι πρέπει να έχουμε μία καταβολή τελών, αλλά τότε θα είναι υψηλό το τέλος. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μια οργανισμός ο οποίος βασίζεται σε επιδοτήσεις. Θέλουμε επί τη βάση της αρχής του οριπέρων πληρώνει να μπορούμε να αντλούμε έσοδα από τις πληρωμές αυτές. Έχουμε βέβαια και κάποιες άλλες πηγές εσόδων γιατί κάνουμε και πράγματα για την Κομισιόν και αξιολογώντας διάφορα προϊόντα. Αυτά είναι λοιπόν κάποιες από τις επιθυμίες που εγώ θα ήθελα να διατυπώσω προσωπικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ανταλλαγή αυτή απόψε και για τις απαντήσεις σας. Θα μείνουμε σε στενή επαφή μαζί σας στο μέλλον η ΕΚΑ είναι πολύ κοντά στο, στις πολιτικές μας προσδοκίες και στις καρδιές μας. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο Ελσίνκι, σε όλο το προσωπικό σας που συναντήσαμε με την αντιπροσωπεία μας και κάθε επιτυχία για τους επόμενους μήνες και χρόνια. Yeah. Then uh, we continue with uh, Συνεχίζουμε επομένω τώρα με το επόμενο. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο τη ημερήσια διάθεξη. Ανταλλαγή απόψεων με έναν άλλον ε, σημαντικό συνεργάτη μας, Ähm, nebendran, ne? Ja, da. Direkt nebendran. Uh, uh, yeah. Could Martin sit, please? Okay. Uh, he gave me some notes, you know. Okay. Uh. So, dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του κ. Τόμας Λönggren, Χαίρομαι ιδιαίτερος που είσαστε μαζί μας. Ακούσατε λίγο πολύ τι συζητήσαμε με το ΕΚΑ και ε, τώρα είναι η σειρά μας να μας εκθέσετε την κατάσταση ε, που αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Πολύ σημαντική δουλειά σας και τα κάνετε εδώ και 10 χρόνια. Είσαστε ένας θεσμός. Ο ίδιος είσαστε ένας ζωντανός θεσμός. Και φέτος ε, ολοκληρώσετε αυτή τη δεκαετία και θα θέλαμε να ακούσουμε τις εμπειρίες μας, τις εμπειρίες σας και επειδή ολοκληρώνω τη θητεία σας την 31η Δεκεμβρίου του 2010, προφανώς ε, είναι από τις τελευταίες φορές που θα σας έχουμε εδώ μαζί μας. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και ε, βουλευτές, χαίρομαι πραγματικά που είμαι εδώ μαζί σας. Είναι η ένατη φορά νομίζω που είμαι εδώ για να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνήθως στις ανταλλαγές αυτές ε, μιλάω για τις επιδόσεις ε, του οργανισμού και τι κάνουμε καθημερινά. Σήμερα θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά τα επιτεύγματα, αλλά θα ήθελα να μιλήσω λίγο γενικότερα για τα φάρμακα και για τον κανονισμό για τα, που αφορά τα φάρμακα και την γενική περίθαλψη του πληθυσμού. Θα, δούμε ποια είναι η σχέση μας και με το περιβάλλον και τι θα γίνει στο μέλλον όσον αφορά τις διάφορες θεραπείες. Λίγα λόγια όμως για τη λειτουργία του οργανισμού. Η Επιτροπή έκανε μία αξιολόγηση σύμφωνα με την νομοθεσία που αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η έκθεση ε, δημοσιεύτηκε στις αρχές του τρέχοντος έτου. Η Ernst Young έκανε την αξιολόγηση και η έκθεση ε, ε, παρουσιάζει τις επιδόσεις του οργανισμού τα τελευταία δέκα χρόνια όπου ήμουν και ο διευθυντής του οργανισμού, είδαν ε, τις επιδόσεις μας, ε, τις συνέκριναν ε, με βάση τους στόχους που είχε θέσει η νομοθεσία, εξέτασαν την αποτελεσματικότητα του οργανισμού και εξέτασαν την, το κατά πόσον η, τα αποτελέσματά μας ήταν έγκαιρα. Τα αποτελέσματα ήταν λίγο πολύ θετικά, πετύχαμε όλους τους στόχους που είχαν τεθεί και κατέληξε η έκθεση στο γεγονός ότι ο οργανισμός είναι αποτελεσματικός και λίγο πολύ ε, σεβαστήκαμε τις νομοθετικές ε, προδιαγραφές τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω να ξοδέψω πολύ χρόνο για να σας μιλήσω για τον οργανισμό και τις επιδόσεις μας, γιατί πιστεύω ότι η έκθεση της Ernst και Young αντικατοπτρίζει πιστά τις επιδόσεις μας, όχι μόνο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στο Λονδίνο, αλλά και για το ε, Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Δίκτυο, το οποίο έχει δημιουργηθεί και τα εθνικά εργαστήρια δηλαδή, τα οποία συνεργάζονται μαζί μας. Λοιπόν, επομένως, ο Οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός είναι σε καλή υγεία αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στα θέματα τα μελλοντικά. Τέσσερα είναι τα βασικά θέματα, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν, ε, ρυθμίζονται τα, ρυθμίζονται το τομέα των φαρμάκων στο μέλλον. Το ένα είναι η παγκοσμιοποίηση της φαρμακευτικής αγοράς, Ολοένα και, πιο, ολοένα και περισσότερο φάρμακα παράγονται και τα ενεργειακή ενεργές ουσίες και το τελικό προϊόν, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις Ηνωμένε Πολιτείες ως συνήθως, αλλά παράγονται στην Κίνα, στην Ινδία κτλ. Επίσης, η έρευνα και η ανάπτυξη των φαρμάκων και των προϊόντων γίνεται σε άλλα μέρη και βλέπουμε ότι πολλές φορές Πολλές από τις κλινικές ε, ε, δοκιμές ε, που θα έοφυλα να γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουν χώρα στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ινδία, στην Κίνα, στην Ελληνική Αμερική. Και αυτό αλλάζει το ρόλο των ρυθμιστών που είμαστε εμείς διότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα όσα γίνονται και σε άλλα εδάφη και διαπιστώσαμε ότι τα προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμίσουμε και να ελέγχουμε ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά δεν ε, παράγονται στην, ε, στο έδαφος μας πλέον. Άρα έπρεπε να λειτουργήσουμε σε μια παγκόσμια κλίμακα, να συνεργαστούμε με άλλους ρυθμιστές στην Κίνα, στην Ινδία παραδείγματο χάρη και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι παίρνουμε όλες τις πληροφορίε σχετικά με την ασφάλεια αυτών των προϊόντων, ε, ε, πληροφορίες ε, για τον κατασκευαστή κτλ. Αυτό είναι, είναι μια νέα πρόκληση για μας και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον σχεδιασμό της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και για το μέλλον. Ότι πρέπει να είμαστε πιο σφαιρικοί έχουμε ξεκινήσει σε αυτό το δρόμο και η Κομισιό έχει λάβει αυτό το θέμα υπόψη της στην πρόταση που έκανε για τα πλαστά φάρμακα. Επομένως υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες από πλευράς της Κομισιό και από πλευράς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να είμαστε ευέλικτοι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σε παγκόσμιο επίπεδο ένα, αυτό, ένα στοιχείο είναι αυτό που μας επηρεάζει. Το δεύτερο είναι οι επιστημονικές εξελίξεις. Τεράστια πρόοδος όσον αφορά τις επιστημονικές εξελίξεις. Νέες ευκαιρίες, νέες θεραπείες. Έχουμε τα, τη γονιδιακή θεραπεία, την κυταρική θεραπεία, τα, οι βιοδείκτες, στοιχεία που αφορούν την γενετική ιατρική. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας ατομικά πλέον τους ασθενείς, ασθενείς που αντιδρούν, ασθενούς, ασθενείς που δεν αντιδρούν. Μπορούμε να παράγουμε νέους ιστούς φοβερές εξελίξεις. Ε. Όμως αυτές οι εξελίξεις ε, πρέπει να επιταχυνθούν και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι θα πρέπει να εκπονήσουμε όλους τους ε, νομοθετικούς κανόνες για αυτά τα νέα φάρμακα τα οποία θα κυκλοφορήσουν στην αγορά. Και νομίζω όμως ότι όλα αυτά έχουν αλλάξει την όλη φαρμακευτική οικολογική αντιμετώπιση για τα νέα φάρμακα, για τις νέες θεραπείες. Ε, θα πρέπει να είμαστε πιο, να δρούμε προληπτικά έτσι ώστε να μην ε, εμφανίζονται ασθένειες. Πρέπει να είμαστε πιο επιλεκτικοί για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι ε, στην επιλογή των φαρμάκων που θα χρησιμοποιήσουμε σε συγκεκριμένους ασθενείς. Νομίζω ότι το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε είναι είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές τις εξελίξεις. Το ε, σύστημα περίθαλψης, ε, το υγειονομικό σύστημα περίθαλψης των κρατών μελών είναι προετοιμασμένο για αυτού του είδους τις εξελίξεις. Ε, μετά υπάρχει αυτό το κανονιστικό χάσμα, πώς το χαρακτηρίζω. Μέχρι τώρα είχαμε ένα σύστημα ευρωπαϊκής έγκρισης, ευρωπαϊκό σύστημα έγκρισης. Γινόταν μία αίτηση, γινόταν μία αξιολόγηση και εδίδοντο μία έγκριση που ίσχυε και στις 27, στα κράτη-μέλη και ο ασθενής είχε πρόσβαση στο φάρμακο. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Οι εθνικές αρχές, οι εξετάζουν ε, την, ε, αποτελεσμα... θα εξετάζουν την αποτελεσματικότητα ε, από πλευράς οφέλους και κόστους για, το... για, κάθε... για κάθε φάρμακο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες εξελίξεις, διότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα σε αυτά τα οποία εμείς σαν αριθμιστές κάνουμε, αλλά και ανάμεσα σε αυτά που 27 κράτη-μέλη ε, κάνουν από την άλλη. Οι 27, κράτη, 27 ε, εθνικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την υγειονομική περίθαλψη. Το πρόβλημα είναι βέβαια να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, γιατί αυτό θα κοστίσει πολλά χρήματα στο μέλλον. Τέταρτος τομέας ε, ραγδαίων εξελίξεων είναι ο τομέας της διαφάνειας. Εάν υπάρχει κάποιος ε, τομέας στον οποίο θα ήθελα να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτά τα 10 χρόνια που, που ήμουνα, που υπηρέτησε τον οργανισμό αυτό, είναι η διαφάνεια και το προσπάθησα αυτό. Αλλά εάν δείτε κανονιστικούς οργανισμούς σαν τον δικό μας σε κάποιον άλλον, δεν είναι εύκολο να είμαστε διαφανείς, διότι από τη μία πλευρά είναι, υπάρχει το θέμα του απόρριτου και από πλευράς βιομηχανίας, μετά είναι το απόρριτο όσον αφορά τα στοιχεία που αφορούν τον ασθενή και μετά βέβαια προφανώς επιβάλλεται η διαφάνεια όσον αφορά την νομοθεσία που θα εφαρμόσουμε. Τώρα, δημοσιεύουμε περισσότερες πληροφορίες, όλο είναι και περισσότερες πληροφορίες. Οι πληροφορίες όμως που έχουμε είναι εκατομμύρια έγγραφα και για να βρούμε ποια είναι το επαγγελματικό απόρριτο, το εμπορικό απόρριτο, ποια είναι τα στοιχεία των ασθενών κτλ. Ε, πρέπει να περάσει πολύς χρόνος, δηλαδή ένα μήνα ένα άτομο μπορεί να ασχοληθεί για να δει κατά πόσο μπορεί να δημοσιεύσει μια πληροφορία ή όχι. Υπάρχει μια νέα απόφαση σχετικά με τη διαφάνεια, θα προχωρήσουμε. Ελήφθη η απόφαση αυτή πρόσφατα Δηλαδή θα δημοσιεύουμε περισσότερες πληροφορίες μένα, όμως θα πρέπει να ρυθμίσουμε καλύτερα και την ροή των πληροφοριών που παίρνουμε. Έτσι ώστε όταν ε, οι πληροφορίες μπαίνουν στο, στον οργανισμό μας να ξέρουμε κατά πόσο μπορούν να δημοσιευθούν ή όχι. Βέβαια επαναλαμβάνω ότι για να είμαστε πλήρως διαφανείς θα μας πάρει πολύ χρόνο. Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικής, βασικοί τομείς που θα επηρεάσουν το φαρμακευτικό περιβάλλον στο μέλλον. Και δεν αφορούν μόνο το, το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αλλά γενικότερα το όλο τοπίο υγείας. Τώρα, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τα φάρμακα και, γενικό, και για το γενικότερα ε, συστήματα ασφάλειας, ε, υγειονομικής ε, προστασίας της υγείας. την φαρμακευτική έρευνα δίδονται πάρα πολλά χρήματα, 80 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Όμως 10 μόρια βγαίνουν κάθε χρόνο. Από αυτά τα μόρια τα οποία, που βγαίνουν, τα οποία βγαίνουν ε, από αυτή την έρευνα. Λίγα είναι αυτά τα οποία είναι όντως ε, θεραπευτικά, αν θέλετε, μπορούν να χρησιμεύσουν ε, στις θεραπείες μετά από έρευνες. Επομένως, αποδίδει η φαρμακευτική έρευνα λίγα πράγματα. Πολλά χρήματα δαπανώνται, λίγα αποτελέσματα, πενιχρά αποτελέσματα έχουμε. Τώρα, στα θέματα των κλινικών ε, δοκιμών. Όταν θέλουμε να εγκρίνουμε ένα φαρμακευτικό προϊόν. Ξέρουμε ότι η αποτελεσματικότητα του προϊόντος ορίζεται σαφέστατα. Υπάρχει όμως και άλλη μια κατάσταση όταν το προϊόν αυτό γίνεται μια πραγματικότητα, μια φαρμακευτική πραγματικότητα. Και το πρόβλημα είναι ότι μπορεί ένα φάρμακο να μην χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των κλινικών ερευνών μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι σύμφωνα με την σήμανση ή χωρίς σήμανση και προφανώς εκεί το όφελος από το φάρμακο αυτό περιορίζεται. Και ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δεν γίνεται μια ορθολογική χρήση των φαρμάκων στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Σε πολλές ε, ε, έρευνες που κάνουμε, μελέτες που κάνουμε, για κάποια φάρμακα όπως το ακόμπλιο παραδείγματος χάρη δεν είναι γιατί μειώθηκε το όφελος του φαρμάκου αλλά γιατί δεν το χρησιμοποίησαν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σωστά. Επομένως, εμείς οι ρυθμιστές, οι νομοθέτες, έχουμε λίγα στοιχεία στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ε, την ορθολογική χρήση των φαρμάκων στην αγορά. στην νομοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα να ε, εκδώσουμε ένα πρόγραμμα ε, περιορισμού των ε, κινδύνων ή της διαχείρισης των κινδύνων. Όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο εάν οι υγειονομικές αρχές δεν το λάβουν υπόψη τους, δεν μπορούν να το εφαρμόσουν αυτό το, αυτή την ελαχιστοποίηση, τον περιορισμό των, των κινδύνων. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα. Δαπανούμε τεράστια ποσά για να βρούμε κάποια φάρμακα και μετά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να, ε, να, να αποδείξουμε ότι χρησιμοποιούνται σωστά τα προϊόντα αυτά, τα φάρμακα αυτά. Και είναι σοβαρό το θέμα γιατί υπάρχουν παρενέργειες από τα φάρμακα κτλ. Επομένως, νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε Βέβαια υπάρχει ελπίδα να είμαστε καλύτεροι, να ε, στοχεύουμε καλύτερα στις θεραπείες με τα φάρμακα. Σήμερα ε, αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο αριθμό ασθενών όπου η απάντηση στα φάρμακα είναι γύρω στο 30%. Άρα τι εννοώ ότι θα πρέπει να δώσεις, να χορηγήσεις το φάρμακο σε 300 άτομα για να έχεις σε 30 άτομα αποτελεσματικότητα. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι 30 δεν το ξέρει κανεί, και κάποιο να χρησιμοποιήσει ένα φάρμακο θέλει να, ή να, να ανήκει σε 30 που θα αντιδράσουν ε, στο φάρμακο. Όμω, η τεχνολογία βοηθάει με αυτού του δείκτε, του βιολογικού δείκτε. και έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε άμεσα τα 30 άτομα τα οποία θα αντιδράσουν στην θεραπεία. Επομένω, στο μέλλον μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, θεραπευτικές ικανότητες των, ε, των φαρμάκων κλιμάκων. αυτό που χρειάζεται είναι επίσης να βελτιώσουμε και τους, τους δείκτες αυτούς. Και στην πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα η Κομισιό δίνει πολλά χρήματα για την ε, δημιουργία και την προώθηση των ε, δικτών, των βιολογικών δικτών. Και χρησιμοποιούμε ορισμένες, ορισμένες αυτού ε, αυτούς τους δείκτες έτσι ώστε να επιλέξουμε ή να αποκλείσουμε ας θέλετε ασθενείς ε, από την χορήγηση κάποιων δεδομένων φαρμάκων και με τον τρόπο αυτό βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Επομένως, στο μέλλον θα πρέπει να στοχεύουμε περισσότερο την χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων και, και θα πρέπει όμως τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ε, να ε, φροντίσουν να βελτιώσουν και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Τι μπορεί να γίνει, πολλά μπορεί να γίνουν. Μία ε, μια πρωτοβουλία ας πούμε αν θέλετε είναι η ενημέρωση των ασθενών διότι ε, οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για, την, ε, για το ενδυνάμει όφελος και αποτελεσματικότητα των φαρμάκων που παίρνουν. Τέλος, όλες αυτές οι πτυχές εξετάστηκαν, τις λάβαμε υπόψη μας και είδαμε τι μπορούμε εμείς σαν ε, οργανισμός να κάνουμε και αυτό έχει συμπεριληφθεί στον ε, οδικό χάρτη της, του οργανισμού και υπήρξε και μία απάντηση πολύ σημαντική από όλους τους ε, ενδιαφερομένους από όλους τους συνεργάτες μας σε τρεις τομείς εμείς έχουμε εστιάσει την προσοχή μας. Το ένα είναι οι ανάγκες της δημόσιας υγείας, ενθαρρύνοντας την έρευνα ε, για παραγωνισμένες και ξεχασμένες ασθένειες. Ε, θέλουμε επίσης να προετοιμάσουμε σχέδια προστασίας του κοινού. Δεύτερον, ε, να βελτιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και να βελτιώσουμε το μοντέλο του οργανισμού όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων ε, των φαρμάκων. Και τρίτος τομέας είναι να βελτιστοποιήσουμε την ορθολογική χρήση των φαρμάκων θα πρέπει να εφαρμόσουμε θέματα φαρμακολογικής ε, επίβλεψης αν θέλετε και θα πρέπει να χορηγούνται πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα τα οποία έχει αξιολογήσει ο οργανισμός Η φαρμακολογική επίβλεψη έχει προβλέψει πολλά νέα εργαλεία τα οποία μας ε, βοηθάνε. Λοιπόν, μετά από αυτή την ε, δημόσια διαβούλευση, ελπίζω ότι θα έχουμε μια, ένα σαφή προσανατολισμό για τον οργανισμό τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για μένα γιατί εγώ φεύγω, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και αυτή την Επιτροπή για την ε, υποστήριξη προς τον οργανισμό, αλλά και για, όλον τον επικοδομη... και για όλη την επικοδομητική κριτική που ασκήσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο την έχετε εσείς κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Λένγκρεν. για την παρουσίαση που μας έκανε. Οι απόψει σας όσον αφορά την μελλοντική αγορά φαρμάκων είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Έχουμε την παγκοσμιοποίηση, την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Μας μιλήσατε για κόστος και την αναγκαιότητα να είναι κανείς συνειδητοποιημένος ε, για το πώς ακριβώς έχει το όλο θέμα να ξέρετε ε, οι απόψεις σας, αυτές οι παρατηρήσεις σας θα ληφθούν υπόψη. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Ε, εδώ έχουμε την Ροντ Μπέρεντ, η οποία ίσως είχατε ήδη την ευκαιρία να αντιμετωπίσετε και κάποιες δυναμικές ε, ε, απόψεις ίσως. Ροντ Μπέρεντ. Ε, ο κύριος Τόμας Λένγκρεν θεωρεί ότι οι υπόψει μας είναι επικοδομητικές. Όπως και να έχει το θέμα, θα ήθελα να πω, οι προτάσεις που γίνατε, οι οποίες δεν ήταν δικές μου, ήταν του Κοινοβουλίου καταρχήν. Πιστεύω, ε, ο κύριος Τόμας Λένγκρεν θεωρεί ότι αυτές οι προτάσεις ήταν θετικέ. Ε, γίνανε, συνετάχθησαν με τέτοιο τρόπο που να φαίνονται σαν είναι δικέ του ίδιε οι ιδέε. δεν θέλουμε μια νέα επιτροπή και για, από τη, για προϊόντα, φάρμακα τα οποία θα είναι παραδοσιακά. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσει κανείς το θέμα μεγάλη πεποίθηση και χαιρόμαστε που έχουμε και την παρουσία εδώ ενός μέλους του Συμβουλίου της Δικήσεως της Υπηρεσίας και χαιρόμαστε για την, αυτή την παρουσία. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η, η παρουσία σας ήταν σημαντική, επικοδομητική και έγινε μια σωστή αγαστή συνεργασία. Χαίρομαι λοιπόν για το έργο το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα. I don't want to put many questions to, to Thomas. In fact, I only want to underline... Είχα να πω απλώς κύριε Λένγκρεν ότι ε, δεν θέλω να σας κουράσω με ερωτήσεις. Γίνατε οι δηλώσεις πραγματικά ενός ε, ε μεγάλου πολιτικού άνδρα. παρόλο που μας είπατε ότι θα, μετά από αυτό εδώ το, το έργο που ολοκληρώνεται θα αποχωρήσετε, θα αφήσετε την υπηρεσία. Για μας να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να, για όλες τις pharmaceuticals which are only for a very small group, if not even only one or two people in the European Union. That will be για όλους εμάς ε, υπάρχει μεγάλη σημασία όσον αφορά τις διάφορες πτυχές, πτυχές που αναγκαστικά δεν είναι μέρος του ε, πεδίου εφαρμογής της υπηρεσίας αυτής. Είναι μια πολύ σωστή προσέγγιση και χαίρομαι που εσείς μιλήσατε για μια αρθολογική χρήση του συστήματος περίθαλψης. Αλλά εμείς εφιστούμε την προσοχή. Ε, ε, έχετε ένα συγκεκριμένο ρόλο σε αυτήν την υπηρεσία σας. Γιατί δεν βρίσκεται μέσα. Μην έχει την ίδια πίεση που έχουν τα κράτη-μέλη, γιατί πολλές φορές η όλη πολιτική για τα φαρμακευτικά συσκευάσματα ακολουθείται από μία πτυχή μονάχα οικονομική και προϋπολογισμού. Και πολλές φορές καταμετράται το οικονομικό κόστος της παράτασης της ζωής ενός ασθενούς. Δεν πρέπει να βλέπουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Η ορθολογική αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι τελείως διαφορετική η δική σας από ότι 27 εθνικών φορέων όπου η πίεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ασφικτική. Και στην Γερμανία έχουμε τέτοια προβλήματα όπου έχει ουσιαστικά ευνοχιστεί η η υγειονομική περίθαλψη από τις πιέσεις των Υπουργών Οικονομικών. Μας ενδιαφέρει επίσης η έρευνα για τους βιο... Ε, για τις ουσίες οι οποίες παίζουν το ρόλο των ε, βιοανιχνευτών. Και αυτό μας ενδιαφέρει όταν έχουμε τις φαρμακευτικές ουσίες, όταν θέλουμε να θεραπεύσουμε ορισμένες ασθένειε και εγώ μιλώ ως νομομαθής δεν είμαι ειδικό στα φαρμακευτικά θέματα, αλλά όταν μιλάμε για οι άσημες ασθένειες, πάντα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους, ε, τις ουσίες οι οποίες είναι βιοσημανσιακές κατά κάποιο τρόπο που δίνουν μια βιοσήμανση στην κατάσταση ορισμένων ασθενειών και που μας βοηθούν να έχουμε μια εξειδικευμένη ως προς το γονιδίωμα μεταχείριση με φάρμακα είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Και φυσικά και η θεραπεία είναι πολύ σημαντική, η εστίασή σας είναι πολύ σωστή. Και τέλος για τις διαφάνειες, Γιατί διαφάνεια μάλλον. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό και ξέρω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων στην αίμα όπως και σε άλλους φορείς Κάτι αντίστοιχο είπα και στον ε, κύριο Ντάνσερ της ΕΚΑ. Η αίμα είναι ίσως σε λίγο καλύτερη κατάσταση γιατί πολύ συχνά οι εμπειρογνώμονες είναι επιστήμονες από εθνικούς φορείς ή από πανεπιστήμια που έχουν ε, μια πιο άνετη κατάσταση αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η αίμα κάνει ανεξάρτητες συστάσεις. Το μας τελειώνω. Όπως είπε και ο κύριος Λάινεν, μπορεί να είναι η τελευταία σας επίσκεψη εδώ εγώ πρέπει να εκφράσω μια πλήρη ευγνωμοσύνη γιατί έχετε καταφέρει να σημαδέψετε την εργασία της ΕΜΑ τα τελευταία 15 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε παίξει και εμείς κάποιο ρόλο στην ε, διαμόρφωση της ΕΜΑ με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ο κ. Νασάουρ. Πολλές συζητήσεις είχαμε που δεν ήταν πάντα εύκολες και ανέμελες. Δεν συμφωνούσαμε πάντα αλλά όσοι βλέπουν σήμερα την αίμα πρέπει να σας επενέσουν για το έργο σας, για τη σωστή σας προσέγγιση, για την σκανδιναβική ομή και σαφή και αντιρομαντική προσέγγιση που αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το οποίο προέχει. Αυτά ήθελα να πω Πάντα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ο Τόμα Λάντμπεν είναι αυτός ο στον οποίο οφείλονται όλα αυτά τα θετικά στοιχεία στην αίμα και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία ξέρουν ότι αυτό που κάνατε μέσα στην ε, αίμα και έναντι του έξω κόσμου ήταν πραγματικά εξαιρετικά αξιέπαινο. Yeah, Ευχαριστώ Δάγμαρ. Ίσως μπορούμε να κάνουμε ένα ποτό μαζί στο μπαρ και εκεί μπορείς να δώσεις στον τόμα όλα τα λουλούδια που έχεις κρύψει σε κάποια γωνιά της αίθουσας. Καθηγητά Λέμαλ, θέλω να σας ε, χαιρετήσω. Είσαστε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και νομίζω ότι θα θέλατε να πείτε κάτι. Αλλά προηγουμένως έχουμε την κυρία Μακέβεν που είναι εισηγήτρια για την φάρμακο επαγρύπνηση. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ. Την ΕΜΑ για την, ΕΜΑ για την δουλειά που έχει κάνει. Όντω ε, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μας έδωσε πολλέ πληροφορίε για, την, ε, για, την, για τα κείμενα αυτά τα οποία ε, υιοθετήσαμε με μια πρώτη ανάγνωση δεν πρόκειται να ζητήσω από ότι όπως και η Ντάγμαρα, τεχνο, τεχνικές πληροφορίες. Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και με τους συνεργάτες σας. Αλλά η πραγματική ζωή, η πραγματική χρήση των φαρμάκων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η ΕΜΑ δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να, να είναι σίγουροι ότι τα φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά είναι ασφαλή. Αλλά θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν, ε, ότι υπάρχουν και οι ασθενείς οι οποίοι πρέπει να ε, παίρνουν κάποια φάρμακα, οι γιατροί θα πρέπει να ξέρουν πώς μπορούν να συνδυάσουν όλα αυτά τα φάρμακα τα οποία είναι απαραίτητα για κάποιον ασθενή κτλ. Μίλησα με έναν εμπειρογνώμονα πριν από μερικές μήνες από το Συνωμένες Πολιτείες και μου είπαν ότι δαπανούν ένα τεράστιο ποσό, μάλλον ένα τεράστιο ποσοστό ε, των φαρμάκων ε, και των χρημάτων ε, για τα φάρμακα στους τελευταίους έξι μήνες της ζωής ενός ασθενούς. Δεν γίνεται μια αρθολογική χρήση των φαρμάκων. Επειδή ξέρουν ότι είναι ετοιμοθάνατος ο, ο, ο ασθενής, του δίνουν ένα σωρό φάρμακα. Δηλαδή γίνονται τεράστιες επενδύσεις χωρίς να, να έχουν να πάρουν και τίποτα πίσω ας πούμε. Και γενικότερα, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ε, ότι όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δίνονται στις φαρμακευτικές εταιρείες ε, θα δόχουν και κάποιο αποτέλεσμα. Ίσως θα πρέπει να έχουμε πιο εστιασμένα φάρμακα. δείτε τι γίνεται με την, ας πούμε, θα μπορούσαμε να ε, συνδυάσουμε την διατροφή και το Alzheimer. Ε, δεν έχει γίνει έρευνα, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει μια έρευνα για, το, για τον τρόπο ζωής του καθενός και την υγεία και τα, τα φάρμακα. Τέλος πάντων, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες αυτές οι έρευνες θα αποδώσουν και κάτι. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις, για τις οποίες ξέρω την απάντηση βέβαια, αλλά απλώς έτσι... Ε, αλλά θα ήθελα, ας πούμε, να, να, να λάβουμε υπόψη μας κάποια πράγματα και κυρίως για την διαφάνεια. Είδαμε τι έγινε με την πανδημία για τη, της σε πέρυσι. Ε, εσείς έχετε πληροφορίες όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, ε, τι πληροφορίες ε, έχετε. Επίσης τα χρήματα που, παίρν, που εισπράτετε από τα τέλη τέλος πάντων. Πολλοί συνάδελφοι είναι εδώ τα τελευταία 15 μήνες και κυκλοφορούν διάφορες πληροφορίες οι οποίες δεν είναι όλες σωστές. Επομένως, καλό θα είναι να γνωρίζουμε όλοι, να γνωρίζει το κοινό ε, κάποιες πληροφορίες. Π.χ. ας πούμε πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα τα οποία εισπράτεται. Ε, ευχαριστώ Λίντα. Χάσατε τη συζήτηση σήμερα το πρωί για την γρήπη ή τα έναν ή ένα. Η Φρανσουάς Γκροστέτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα φυσικά να απευθυνθώ στον διευθυντή μας λέγοντάς το ότι 10 χρόνια που πέρασε επικεφαλής της ΕΚΟΦ ε, ήταν χρόνια ανάπτυξης της υπηρεσίας. Ανάπτυξη η οποία αναγνωρίζεται από όλους. Είναι και η αξιοπιστία που δημιουργεί το οποίο δεν ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκέ υπηρεσίε. Πραγματικά σας συγχαίρω για το έργο σας επικεφαλής αυτής της υπηρεσίας. Επίσης, να, όπως είπε και η Ντάγμαρ, να πω ότι εγώ εκτίμησα ε, την ε, σκανδιναβική σας έλεγα αυστηρότητα, η οποία οδήγησε μια κατάσταση, ε, μαζί σας, δημιουργήθηκε μια εμπιστοσύνη Μα δίνατε τακτικά ε, πληροφορίες. Αυτό ήταν σημαντικό, το επαναλαμβάνω, ότι ειλικρινά υπάρχουν τόσα και τόσα που μπορούν να λεχθούν και πολλέ φορές υπάρχει παραπληροφόρηση, ξέρετε. Εδώ, στο Κοινοβούλιο, εδώ, σε συνάντηση με εσά, εμείς είμαστε ε, σε μια επαφή για να δουλέψουμε για το γενικό συμφέρον, για να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη της υγείας. Αυτό είναι βασικό. Και αν πιστεύουμε ότι μπορεί να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε αυτή την Ευρώπη της υγείας, αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο συριζόμενοι στην ε, υπηρεσία σας, στο έργο το δικό σας. Ειλικρινά. Ε, υπάρχουν υποψίες ε, όσον αφορά κάποιους εμπειρογνώμονες. Ε, απειλούνται μερικοί από αυτούς από εμά ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων αλλά θα ήθελα να πω βασικά δεν είναι θέμα υποψίας. Εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ αμφιβολίες όσον αφορά το έργο σας, την αυστηρότητα που δείξατε. Σας το παναλαμβάνω, ξανά λέω ευχαριστώ και πραγματικά θα μας λείψετε. Τούτων λεκθέντων να έρθω στο θέμα της αξιολόγησης των τεχνολογιών για την υγεία. Εσείς κάνατε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τη χρήση ε, σε υπηρεσίε εθνικών επίπεδου, η χρήση φαρμάκων τα οποία δεν έχουν την ε, καθαρή έγκριση, ε, θέματα ποσολογίας επίσης. Όλα αυτά είναι σοβαρά. Είπατε, εκφράσατε τους φόβους σας για κάποια φάρμακα για κάποια φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένε περιπτώσει καρκίνου. Αλλά χρησιμοποιούνται στη Μεγάλη Βρετανία Φερρυπίν για οφθαλμολογικά προβλήματα. Πραγματικά υπάρχουν τόσε και τόσε περιπτώσει που δημιουργούν ε, ε, ερωτηματικά και αμφιβολίες. Μας λέτε ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα να διαδράσουμε με τις εθνικές υπηρεσίες πραγματικά θα ήθελα να σα ρωτήσετε στη δράση που θέλετε να κάνετε στα πλαίσια τη υπηρεσία. Έχετε και την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ναι ή όχι. Και πώς σκοπεύετε να αναπτύξετε αυτό το θέμα της ευρωπαϊκής αξιολόγησης των τεχνολογιών που αφορούν την υγεία. Εσείς σύντομα θα εγκαταλείψετε την υπηρεσία, αλλά σίγουρα θα μετα δώσετε την πείρα που έχετε στους ε, ανθρώπους που σας διαδεθούν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, θα δώσουμε το λόγο. Κυρία Ριβάς, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε ότι θέλουμε μια Ευρώπη για την υγεία. Θα ήθελα όμως να πω τα εξής για την ποιότητα της επιστημονικής αξιολόγησης. Για πείτε μου, έχετε κάποιες προτάσεις να κάνετε ούτως ώστε να βελτιωθεί το πρωτόκολλο που αφορά την επιστημονική αξιολόγηση. Για το Ταμιφλού Φερρυπίν, η πολεμική που είχαμε. Γίναν μελέτες, ξέρετε, από το British Medical Journal, όπου λέγανε αυτές οι μελέτες όσον αφορά το ταμιφλού ήταν μελέτες που γίνανε από, ε, από αυτούς που παρήγαγαν το ταμιφλού και το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε ότι έχουμε καλύτερες ε, ε, μελέτες. Συχνά είναι οι χώρες μέλη που κάνουν τις αξιολογήσεις. Δεύτερο ερώτημα. Όσον αφορά την διαδικασία fast track, τι σκοπεύετε να κάνετε θα τη διευρύνετε και σε άλλα φάρμακα ή μήπως για σας είναι μια διαδικασία έκτακτη. Ε, και τέλος, μια τελευταία ερώτηση. Όσον αφορά τις επιπόπτεις ε, των φαρμάκων στο περιβάλλον, διαπιστώνουμε όλο και πιο πολύ ότι υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία είναι πολύ ανθεκτικά, υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον ε, ενισχύονται τα βακτηρίδια, υπάρχουν ενδοκρινολογικές επιπτώσεις. Έχετε λοιπόν τη θέληση στην υπηρεσία σας να λάβετε υπόψη ε, τις επιπτώσεις ε, αυτών των φαρμάκων στο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Παρβάνοβα, δεν μπόρεσα να έρθω προηγουμένως στην ε, συνεδρία σε αυτή και δεν ξέρω αν τέτοιο αυτό το ερώτημα. Θέλω να θέσω όμως το ερώτημα για τον, σε σχέση με τον νέο ρόλο και τα καθήκοντα του φορέα σας που έχουμε προβλέψει στην οδηγία περί φαρμακευτικών και επίσης στην οδηγία κατά των παραποιημένων φαρμάκων. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτά τα διευρυμένα καθήκοντα και μπορούμε εμείς να σας βοηθήσουμε σε χρηματοοικονομικό επίπεδο για να καλύψετε το πρόσθετο κόστος. Και εγώ είχα να κάνω ε, μια ερώτηση σε σχέση με το ερώτημά σας για την ε, χρησιμότητα. Όπως ξέρετε στη Γερμανία αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα μια μεγάλη συζήτηση για την αξιολόγηση των φαρμάκων, τι είναι χρήσιμο, τι δεν είναι χρήσιμο. Αν κατάλαβα σωστά τα, τα νούμερα, η Ελβετία έχει 2.000 συγκεκριμένα φάρμακα και εμείς έχουμε 20.000. Βέβαια είναι πιο μεγάλη αγορά η Γερμανία, αλλά πραγματικά τίθεται σε ευρύτερο επίπεδο το ερώτημα του ποια φάρμακα είναι χρήσιμα και ποια δεν είναι χρήσιμα και λέγεται ότι πολλά από τα φάρμακα, τα καινούρια φάρμακα που έχονται στην αγορά δεν έχουν κάποια προσθέμενη αξία, δεν προσθέτουν, δεν κομίζουν γλάφκα στην Αθήνα ή τουλάχιστον στη Γερμανία. Είναι τα ίδια φάρμακα που είχαν τι παλιέ ενεργέ ουσίες. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχόλια για όλα αυτά τα θέματα και ο καθηγητή Λέμελ επίσης, ο οποίος είναι ο αντιπρόσωπο του Κοινοβουλίου, τι έχετε να πείτε για τα θέματα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου και είμαι πολύ ευτυχή. Και θέλω να πω κάτι επί τη ευκαιρία του, της ε, αποχώρησης του Τόμας, όχι από τον, την εγώ υπηρεσία, αλλά από την διοίκηση της ΕΜΑ. Από το 2001 είναι εκτελεστικός διευθυντής ο Τόμας. Δύο φορές είχε τη θητεία αυτή του Προέδρου του Επικεφαλής Υπηρεσία σε αυτή την τόσο σημαντική και νευραλγική θέση. Το 2001 η ΕΜΑ ήταν έφηβη. Μεγάλωσε και ανδρώθηκε μάλλον γυναικώθηκε με την προεδρία του Τόμας. Ήταν η κινητήρια δύναμη που έφερε την αίμα σε μια από τις πιο προεξάρχουσες θέσεις στον κόσμο και χάρη στην πίεση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργήθηκαν νέες επιτροπές για τα φαρμακευτικά συσκευάσματα για νέε θεραπείε για την ασθενειών όπω ο καρκίνο. Όλε αυτέ οι επιτροπέ πιστεύω ότι χρειάζονται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη να έχουμε μια αποτελεσματική ιατρική για τους λαούς της Ευρώπης. Ως φαρμακολόγος ξέρω ότι πάρα πολλές φορές πολλά αυτά τα φάρμακα που δίνουμε στα παιδιά είναι τρομερά. Δεν το πιστεύει ο άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των φαρμάκων. Υπάρχουν σημαντικέ προκλήσει που θα πρέπει να τύχουν απαντήσεων και ο Τόμα Λάντκριν, ω εκτελεστικό διευθυντή τη ΕΜΑ, νομίζω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική εργασία για να αντιμετωπίσει αυτέ τι προκλήσει. Θα πρέπει όμω να θυμόμαστε ότι ένα αποκεντρωμένο φορέα όπω η ΕΜΑ δεν μπορεί αμέσω πάντα να παίρνει μια απόφαση η οποία είναι ε, από την πρώτη στιγμή η σωστή. Δεν είναι όλες οι αποφάσεις εύκολο να γίνονται δεκτές ομόφωνα από όλους τους εμπλεκομένους και από όλους τους επιστήμονες. Μόλον τούτο, ένας εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και τα αντιμετώπισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να καταλήξει σε απαντήσεις και αποφάσεις. Στην εισαγωγική του ομιλία ο Τόμας αναφέρθηκε στα μελλοντικά προβλήματα αποκλήσεων, ε, παγκοσμιοποίηση, επιστημονικά σώματα, διαφάνεια, αριθμιστική φορείς. Όλα αυτά τα θέματα έχουν συζητηθεί και θα εξακολουθούν να συζητούνται στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Και πραγματικά θα ήθελα να απαντήσω μερικά από τα ερωτήματα Η φαρμακολογία είναι μια επιστήμη που βασίζεται στις πιθανότητες. Δεν είναι μια επιστήμη όπου υπάρχει 100% ασφάλεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η παθοφυσιολογία των ανθρώπων είναι πολύ πολύπλοκη. Θα πρέπει να τα γνωρίσουμε λοιπόν όλα αυτά και παρέχουμε στο δικό σας ερώτημα. Ε, υπάρχουν πάντα όλα αυτά τα στοιχεία, παραγωγικά για τις μελέτες που έχουν γίνει, οι κλινικές μελέτες. Οι κλινικές μελέτες πολλές φορές γίνονται σε εικοσάριδε άντρες, οι οποίοι είναι σε πολύ καλή υγεία. Οι γυναίκες είναι πολύ πολύπλοκες και γι' αυτό δεν τις χρησιμοποιούν στις κλινικές μελέτες. Πρέπει οι κλινικές μελέτες να γίνονται και σε άνδρες και σε γυναίκες. Και έχουμε πια στοιχεία που δείχνουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετικούς κινδύνους και αντιδρούν διαφορετικά στα φάρμακα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν. για τις συγκρούσεις συμφερόντων. Αυτό δεν έχει συζητηθεί ακόμα πλήρως από το Διοικητικό Συμβούλιο, απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι δεν ζούμε σε κενό αέρος. Χρειαζόμαστε εμπειρογνώμονες, χρειαζόμαστε επιστήμονες. Αν βρείτε ένα επιστήμονα ο οποίος δεν έχει κανένα, καμία σύνδεση με την βιομηχανία, δεν είναι επιστήμονας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην διώχνουμε άτομα μόνο και μόνο, μόνο, και μόνο γιατί έχουν κάποια σύνδεση με τις επιχειρήσεις. Το θέμα αυτό της σύγκρουσης συμφερόντων είναι ένα πάρα πολύ λεπτό και δύσκολο σημείο. Μπορούμε να δηλώσουμε όλα αυτά τα οποία κάνει κανείς, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζομαστε στην ΕΜΕΑ, χρειαζόμαστε εμπειρογνώμονες. Τέλος. Ήταν ένας εξαιρετικός εκτελεστικός διευθυντής και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να την συγχαρούμε που τον έθεσε σε αυτή τη θέση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Τόμας για όλα αυτά που έχει κάνει για την Ευρώπη. Λοιπόν, πριν, πριν φύγετε όμως πρέπει να απαντήσετε τα ερωτήματα, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα ευγενικά σας λόγια. Πριν απαντήσω, να ευχαριστήσω και την Dagmar για την υποστήριξη ε, της όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζω να συνεχίσει να υποστηρίζει τον οργανισμό και μετά την αποχώρησή μου. Ευχαριστώ κύριε Γκροστέτ επίσης για όλη την υποστήριξη που μας προσφέρατε όλα αυτά τα χρόνια. Και Λίντα, εσύ είσαι πιο πρόσφατη, αλλά και σε ευχαριστώ για την υποστήριξή σου για αυτό το πακέτο φαρμακοεπίβλεψης, φαρμακοπαρακολούθησης. Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσω να εξηγήσω πώς δημιουργήθηκε αυτό το κανονιστικό πλαίσιο για να μπορέσετε να καταλάβετε τον, το σύστημα αξιολόγησης των ωφελιών των φαρμάκων η βιομηχανία έκανε μέχρι τώρα τις περισσότερες μελέτες. Ε, αυτοί μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ε, τις μελέτες. Αυτό δεν ισχύει στην Ευρώπη μόνο, αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Και στην FTA και στην Κορέα και στην Κίνα και στην Ινδία, σε όλες τις χώρες του κόσμου ε, το βασικό κριτήριο είναι ότι ε, εμείς βάζουμε κάποιες απαιτήσει, η βιομηχανία πρέπει να σεβαστεί αυτά τα κριτήρια και να προχωρήσει σε μελέτες. Οι μελέτες αυτές βέβαια μετά θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης από πλευράς μας ιδιαίτερα κριτικής αξιολόγησης. Τώρα όσον αφορά την χρηματοδότηση των ε, κανονιστικών ε, οργανισμών χρηματοδοτούνται από τα τέλη που πληρώνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, όχι από το δημόσιο. Επομένως, αυτό το οικονομικό μοντέλο δεν το έχουμε μόνο εμείς στην Ευρώπη. Τώρα, το πρόβλημα που τίθεται είναι το εξής. Πώ θα είμαστε σίγουροι ότι τα τέλη αυτά τα οποία πληρώνουν οι φαρμακευτικέ βιομηχανίε δεν θα επηρεάσουν το έργο μα και την αξιολόγηση που κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ προσεκτικά τι κάνουμε, ποιοι είναι οι κανόνε λειτουργίε μα, πώ γίνεται η κατανομή των ευθυνών. Να μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση τα χρήματα τα οποία εισπράττουμε ε, θα επηρεάσουν την απόφαση ε, των αρμοδίων επιτροπών. Ο τρόπος με τον οποίο να δημιουργούμε αυτή την ε, ε, ποιοτική εγγύηση, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ αυστηρός. Ο πλέον αυστηρός από τον κόσμο. Να σε εξηγήσω γιατί. Διότι καταρχάς έχουμε την αίτηση η οποία υποβάλλεται. Αυτή η αίτηση υποβάλλεται στην Επιστημονική ε, Επιτροπή. Αυτή η Επιτροπή έχει έναν εκπρόσωπο ανακράτος μέλος που διορίζεται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εκπροσωπεί δηλαδή αυτός ο άνθρωπος το κράτος μέλος στην Επιτροπή. Όλοι αυτοί μαζί αποφασίζουν να διορίσουν έναν εισηγητή. Και αυτός ο εισηγητής έχει την ευθύνη να αξιολογήσει την ε, αίτηση την οποία έχει υποβάλει η ε, βιομηχανία, η εταιρεία. Και δεν είναι ένας, είναι δύο που ανεξάρτητα ο καθένας κάνει την αξιολόγηση. Και αυτή η αξιολόγηση γίνεται στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, από τις εθνικές υπηρεσίες και μετά τα αποτελέσματα επανέρχονται στην Επιτροπή και συζητώνται και σχολιάζονται κριτικά οι εκθέσεις αυτές από την Επιτροπή, από όλους τους υπόλοιπους εκπροσώπους των 27 κρατών μελών. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι δίνουν ένα feedback στους εισηγητές και γίνεται μια διάφανη και αποδοτική συζήτηση στην, ε, στην Επιτροπή. Απευθύνονται τα ερωτήματα αυτά στην ε, εταιρεία στην, και η, εταιρεία απαντά. Και οι απαντήσεις αυτές αξιολογούνται από τον εισηγητή. Πέραν αυτού του συστήματος έχουμε την ε, peer review team έναν άλλον μηχανισμό δηλαδή που είναι η αξιολόγηση των ομοτήμων και η ομο... έχουμε ανεξάρτητους εισηγητές που σχολιάζουν τις εκθέσεις των πρώτων εισηγητών. Και μετά έχουμε και μία επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή με ανεξάρτητους ε, ε, επιστήμονες τους οποίους, έχουμε, τους οποίους καλούμε και τελικά όλα αυτά υποβάλλονται στην Επιτροπή για την τελική απόφαση και εκεί γίνεται η στάθμιση του κινδύνου και του του ωφέλους. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε μια τέτοια διαδικασία. Είναι μοναδική και πραγματικά μας έχουν δώσει συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Παρόλα αυτά βελτιώνουμε ακόμα περισσότερο τον τρόπο με τον παίρνουμε τι αποφάσει. Διότι η Επιτροπή προσπαθεί να δει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την διαδικασία για την αξιολόγηση του, των κινδύνων και των ωφελιών. Αυτή είναι μια δουλειά που συνεχώς συνεχίζεται έτσι ώστε να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας. Το γεγονός ότι υποβάλλονται τέλη, ε, το ότι πληρώνουν δηλαδή τέλη φαρμακευτικές βιομηχανίες, δεν επηρεάζουν καθόλου τον τρόπο που λειτουργούμε. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Επίσης ήθελα να μιλήσω για το θέμα της διαφάνειας και το έθιξε το θέμα αυτό και στην παρουσίαση που έκανα. Εμείς έχουμε καλές προθέσεις. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, είμαστε όντως διαφανείς. Κάθε εβδομάδα δημοσιεύαμε μία ενημερωμένη έκθεση για τα όλα όσα γινόντουσαν ε, για την φαρμακοεπαγρύπνηση. Τα δημοσιεύαμε στην, στο website μας και ε, δημοσιεύαμε και όλες τις παρενέργειες και όλα τα προβλήματα. Στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου πήραμε μια απόφαση και για την πρόσβαση στα έγγραφα και θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Αυτό τι σημαίνει ότι θα δημοσιεύουμε όλο ένα και περισσότερες πληροφορίες. Θα παίρνουμε αποφάσεις ε, για την δημόσια πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων της φαρμακοεπαγρύπνησης. Θα γίνει μια αναδιάρθρωση, μια αναβάθμιση της τράπεζας δεδομένων για, τις, για τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών, όπου θα καταγράφονται όλες οι κλινικές δοκιμές σε όλη την Ευρώπη και τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών. Επομένως βλέπετε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε περισσότερη διαφάνεια. Πολλά αιτήματα υποβάλλονται στον οργανισμό, όμως πολλά από αυτά τα αιτήματα απαιτούν ε, τη δουλειά ενός ατόμου για πολλούς μήνες για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όλες τις απαραίτητες ε, πληροφορίες. Εάν απαντούσαμε σε όλα τα αιτήματα θα, θα σταματούσε η δραστηριότητα του οργανισμού όμως προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια ροή πληροφόρησης, δηλαδή από να, μπορεί να δημοσιεύεται η πληροφορία τη στιγμή που μπαίνει στον οργανισμό. Εκεί όμως χρειαζόμαστε την βοήθεια της φαρμακοβιομηχανίας για να ξέρουμε ότι μπορούμε να δημοσιεύσουμε κάποιες πληροφορίες. Αμέσως να το ξέρουμε αυτό. Πάντως τώρα όταν είχαμε, όταν είχαμε δημοσιεύσει μια κλινική, τα αποτελέσματα κάποιων κλινικών δοκιμών, ε, ο Ευρωπαίος Ομπούτσμαν ε, μας ε, άσκησε κάποια κριτική, την οποία και λάβαμε υπόψη μας. Τέλος πάντων, όσον αφορά τη σύγκρουση των συμφερόντων. Αυτό το λαμβάναμε ανέκαθεν υπόψη μας. Είχαμε ήδη μια αυστηρή νομοθεσία, ήδη τώρα στη νέα, στο, τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο ενισχύσαμε τις, ε, τις διατάξεις, προσπαθήσαμε να ρυθμίσουμε όλες τις περιπτώσεις ε, ε, σύγκρουση συμφερόντων. Έχουμε ε, επιβάλει υποχρέωση οποιοδήποτε πυρογνώμονες αμέσως να δηλώνει αν έχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων και αν και εφόσον να το δηλώσει θα πρέπει να απομακρυνθεί από την Επιτροπή. Τέλο πάντων, η νέα νομοθεσία, η πιο αυστηρή νομοθεσία θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του επόμενου έτους και με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι θα αλλάξει κάπως και ο τρόπος ε, αντιμετώπισης ε, των περιπτώσεων αυτών. Όμως, όπως είπε ο κ. Λέμερ, δεν μπορεί να έχει εμπειρογνώμονα ο οποίος να μην έχει καμία σχέση με τις φαρμακοβιομηχανίες Δείτε ας πούμε τα θέματα των προηγμένων ε, ε, θεραπείων, ε, κυταρικές θεραπείες, γονιδιακές θεραπείες κτλ. Όλη αυτή η έρευνα χρηματοδοτείται από τις φαρμακοβιομηχανίες. Και αν, πρέπει να, αν θέλουμε να έχουμε μαζί μας αυτούς τους εμπειρογνώμονες, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Όμως, τι αποφασίσαμε για τη σύγκρουση συμφερόνων. Ότι θα διαχειριστούμε το επίπεδο σύγκρουση συμφερόντων και θα διαχειριστούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτή η σύγκρουση να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και τις συμβουλές που δίνουν. Δηλαδή, εάν η συνεισφορά τους δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα, τότε θα την λάβουμε υπόψη μας. Με αυτόν τον τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Και αυτού του είδους οι συγκρούσεις συμφερόντων θα δημοσιοποιούνται. Επίσης, άλλο θέμα, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχει τώρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και έχουμε ξεκινήσει τρει δραστηριότητε. Η πρώτη δραστηριότητα είναι ότι έχουμε καλέσει τα σώματα, αν θέλετε, τεχνολογίες της υγείας, φορείς τέλο πάντων, να μας πούνε κατά πόσον υπάρχουν νέα φάρμακα και εάν υπάρχουν απαιτήσει για κάποιες κλινικές δοκιμές και με τον τρόπο αυτό η φαρμακοβιομηχανία δεν χρειάζεται να επαναλάβει τις δοκιμές. Δεύτερον, βελτιώνουμε τις πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στο ΙΠΑ. Ε, επομένως, όλοι αυτοί οι φορείς θα έχουν ε, περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή τους όταν εξετάζουν την, ε, τη σχέση ωφέλους, κόστους και ωφέλους για να, όταν παίρνουν τις τελικές τους αποφάσεις και ελπίζω ότι στους επόμενους μήνες, σε δύο μήνες, θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το ΙΠΑΡ. Τρίτος τομέας είναι τι γίνεται όταν κυκλοφορήσει το φάρμακο. Το παρακολουθούμε στην αγορά. Τώρα με τα σχέδια ε, αξιολόγησης μπορούμε να παρακολουθήσουμε το φάρμακο και την αποτελεσματικότητα του φάρμακου και μπορούμε τα στοιχεία αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς έτσι ώστε να μην ε, γίνονται διπλές μελέτες. Δηλαδή ο στόχος είναι να μην, γίνονται, ε, να μην γίνεται διπλή δουλειά. Και δηλαδή να χρησιμοποιούμε όσα γίνονται πριν δοθεί η έγκριση και ε, για μετά την χορήγηση της έγκρισης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσον χρειάζεται ε, η μία δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την τεχνολογία και την ορολογία κτλ εφόσον ορισμένα πράγματα γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν χρειάζεται να γίνουν και σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια, για να γίνει κατέληξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να, υιοθετη... να ληφθεί μια πολιτική απόφαση. Πρέπει να υπάρχει πολιτική θέληση. εάν γίνει η αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άκουσα τον πρόεδρο ότι, της Επιτροπής ότι θα κάνει κάποιες δηλώσεις ε, και, ε, ε, για τις προθέσεις της Κομισιόν την επόμενη χρονιά, αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει στο μέλλον. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ όσον αφορά τις δραστηριότητε του οργανισμού. Θα πρέπει βέβαια Α, ξέχασα κάτι. Θα πρέπει να, να, να, να απαντήσω για το ταμιφλού. Ενδιαφέρον θέμα. Ο συνήθως, όταν αξιολογούμε τα, τα φάρμακα, έχουμε πολλές μελέτες στη διάθεσή μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Επιτροπή το εξετάζει, όλε αυτές τις μελέτες. Όταν ένα φάρμακο κυκλοφορεί, μα ε, ε, μας υποβάλλονται μελέτες, αποτελέσματα κτλ και τα αποτελέσματα πολλές φορές των μελετών είναι ε, αμφιλεγόμενα. Γι' αυτό θα πρέπει να αξιολογούμε συνέχεια τις μελέτες και να δούμε κατά πόσον οι μελέτες αυτές είναι σωστές και να δούμε κατά πόσον οι μελέτες αυτές απαντούν και στα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει εμείς. Και πολλές φορές είπα ότι οι μελέτες μπορεί να είναι συγκρουόμενες και να είναι αμφιλεγόμενες. Τελικά όμως η Επιτροπή αυτό το οποίο θα κάνει είναι μια σφαιρική αξιολόγηση. Η μελέτη παρουσιάζει κάποια κενά, κάποια ε, προβλήματα και θα πρέπει να συνδυάσουμε όλες τις μελέτες έτσι ώστε να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό έγινε και για το Ταμιφλού. Και μπορώ να σας πω ότι η Επιτροπή πιστεύει ακόμα ότι η σχέση ωφέλους ε, και κινδύνου για το ταμιφλού είναι θετική. Για το, για το ταμιφλού έχουν γίνει πολλές μελέτες, άλλες θετικές, άλλες αρνητικές και προσπαθούμε να κάνουμε ε, μια αξιολόγηση της κάθε μελέτης και η Επιτροπή μας είναι αρμόδια πάνω στο θέμα. Γιατί έχουν τις τους καλύτερους εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή και εγώ τους έχω εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λέντρε. Νομίζω ότι και εγώ εξ ονόματος όλης της Επιτροπής μας μπορούμε να σας, ευχαριστήσω για την θαυμάσια σας εργασία και να επιβεβαίωσω αυτά τα οποία έπανε οι συνάδελφοι την κυρία Ρότμπερα την ξέρετε εδώ και 10 χρόνια την κυρία Γκροστέτ επίσης εγώ έχω παρακολουθήσει επίσης πρόσφατα τα θέματα αυτά και σίγουρα η οφορέας του Λονδίνου είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για τη διαδικασία έγκρισης των φαρμάκων και ανταποκρίνεται στις ψηλέ προδιαγραφές που θέτουμε πάντα σε τέτοιους φορείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λέντγκρεν. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες που έχετε μαζί σας. Νομίζω ότι από ό,τι έχω ακούσει έχετε και ταλέντο σκανδιναβικό και στο γκολφ και επομένως μπορείτε να εφαρμόσετε και εκεί το ταλέντο σας. Αλλά κυρίως θέλω να τονίσω την αναγνώριση που έχουμε όλοι για το έργο σας και φυσικά και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010 θα ενδιαφερόμαστε να έχουμε την πείρα σας, την εμπειρογνωμοσύνη σας για όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ήρθατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω ότι και στο μέλλον θα βοηθήσετε την Επιτροπή μας και θα μας βοηθήσετε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις οι οποίες ε, θα αναδύονται στον τομέα αυτό. Κλείνει λοιπόν η συνεδρίασή μας, στις 22 Νοεμβρίου θα ξαναβρεθούμε και τώρα στις 6 θα συγκεντρωθούν εδώ συντονιστές για την